So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung des Ausschusses. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είμαστε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Μια και από πλευρά τη συναδέλφου ως Προέδρου προηγούμενα μέχρι το 11 φτάσατε και τα κατάφερε η κυρία Λεπάς. Πάμε στο 12, ένα φλέγον θέμα στην ημερήσια διάταξη. Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα είναι το θέμα μας. Ένα θέμα που ήδη στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία είχαμε εξετάσει με πάρα πολλές τροπολογίες, πάμπολες τροπολογίες των μελών. Και η κυρία Ρενάτε η συνάδελφος κυρία Ζώμερ, ήδη τότε είχε αναλάβει αυτή την έκθεση και έχει και τώρα αυτή την έκθεση. Έχει εμβαθύνει πολύ στη μελέτη αυτών των θεμάτων η συνάδελφος Ζώμερ και της δίνω τον λόγο να μας τα εξηγήσει, να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία που μπορεί κανείς να αποκομίσει για την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα. Κυρία Ζόμερ, έχετε τον λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος φάκελος αυτός που απομένει να εξετάσουμε. Ο Πρόεδρος το είπε ήδη κατά τα τέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Είχα αναλάβει έκθεση για αυτό το χαρτοφυλάκιο, το, την οποία είχα συντάξει. Κατατέθηκαν όμως τόσο πολλές τροπολογίες, χίλιες ε, 332 το καλοκαίρι, σύντομα πριν από τις ευρωεκλογέ, ώστε αποφάσισε η κοινοβουλευτική μας επιτροπή το χατοφυλάκιο να το αναβάλει προς εξέταση στη νέα κοινοβουλευτική θητεία. Η εντολή μου ήταν να ξανασυντάξω την έκθεση για τη νέα θητεία και να προσπαθήσω όσον αφορά τις τροπολογίες τις το δυνατόν περισσότερες να τις ενσωματώσω σε αυτή τη νέα μου έκθεση. Αυτό οδήγησε φυσικά στο από πλευράς όγκου να έχει αυξηθεί η έκθεσή μου εν μεταξύ. 201 τροπολογίες ε, που προτάθηκαν και πραγματικά πολύ ε, ευσυνείδητα επεξεργάστηκαν τις τροπολογίες, όμως ωστόσο θα το κατανοήσετε αυτό, παρέμεινα πιστή στη δική μου γραμμή πλεύσης αρχικά από πλευρά ουσία, από τον μύτο τη Αριάδνη, την πορεία που ακολουθούσε η έκθεσή μου, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να επισέλθω σε κάθε λεπτομέρεια. Μπορώ όμω να σα πω ότι έχει πολλέ λεπτομέρειε η έκθεσή μου πρέπει να εμβαθύνεται σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όσοι είναι παλαιότεροι το κάνανε αυτό ήδη και έχουν εξοικειωθεί με αυτές τις λεπτομέρειες στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. 53 άρθρα και 53 παραρτήματα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα αυτά συνδέονται και είναι συνειφασμένα πολύ στενά μεταξύ τους. Αν δείτε ποιες επιπτώσεις έχει αυτό η μία πρόταση σε ένα άρθρο ή σε παρατήματα ή όπου και περαιτέρω τροπολογίες χρειάζονται για να ρυθμιστούν κάποια πράγματα, προσπαθήσαμε να είμαστε συνεκτικοί και περιεκτικοί. Και ευθύ εξ αρχή πρέπει να ε, καταγγείλω κάτι, να στυλιτεύσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε ένα τόσο τεράστιο εύρος κατέληξε όπου το σύνολο των τροφίμων σε, στα 27 κράτη-μέλη αφορώνται άμεσα τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ κακή αυτή η πρόταση ο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν σκεφτώ πόσοι άνθρωποι είναι ω στελέχη στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συντάξουν ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο και εδώ με ποιους ισχνούς πόρους απίστευτα απαράδεκτους εργαζόμαστε εμείς στην Ευρωβουλή για να αντισταθμίσουμε τα λάθη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα βιώσιμο, πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά ανέσχυντο αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πραγματικά ξεδιάντροπη. Αλλά πρέπει να το πω αυτό έτσι ρητά και κατηγορηματικά για ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο και για πολλά πράγματα που έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και δεν είναι ρεαλιστικά, τα απορρίπτουμε. Και η ίδια η Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στην εντολή τη και δεν κάνει τη δουλειά τη. Αυτό ο νέο κανονισμό θέλει να εναρμονίσει στην ενιαία εσωτερική αγορά, τη νομική ασφάλεια για τους παραγωγούς τροφίμων και τους εμπόρους θα, θέλει, θα έπρεπε να την ε, βεβαιώνει, να την ε, ενισχύει. Θα έπρεπε να αποσυμφορήσει το γραφειοκρατικό βάρος. Σε κανένα από αυτά τα σημεία δεν ανταποκρίνεται το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό έχουμε τεράστια δουλειά ως Ευρωκοινοβούλιο και ξέρω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς εργαζόμαστε έντονα και με μεγάλη, μεγάλο συνέστημα ευθύνης και γνωρίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό σας προσκαλώ να ασχοληθείτε με αυτό το χαρτοφυλάκι. Είναι πολύ σημαντικό και πολλά πράγματα εξαρτώνται από αυτό. Θέλω να υπενθυμίσω για εκείνους που δεν το γνωρίζουν, ο στον των τροφίμων στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που εμπλέκονται. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά πάνω από το 80% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πάμε και σε βιοτέχνες, χειροτέχνες, ε, μικροφουρνάριδες, ε, μικρομαγαζιά. Αυτά όσον αφορά το κείμενο για κάθε επιχείρηση πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Δεν πρέπει να κλείνουν κάποιε επιχειρήσει επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποιου όρου και προποθέσει και η επισήμανση, η ετικέτα για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ταιριαστή σε κάθε ε, προϊόν που αφορά εδόδημο είδο, τρόφιμα και ε, γι' αυτό προτείνω να έχουμε μία υποχρεωτική βάση επισήμανσης ή ετικετοποίησης σε αυτό το νομοθέτημα. Γιατί διότι έχουμε επιπρόσθετα το πρόβλημα σε σχέση με αυτό το νομοθέτημα ή την πρόταση που ετέθη επί τραπέζης, χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλει ο καταναλωτής, τι θέλει ο καταναλωτής όσον αφορά την ετικετοποίηση τροφίμων, τι κατανοεί, τι ζητάει η μάζα των καταναλωτών στην Ευρώπη για αυτό το θέμα τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να το έχουν με βιώσιμο τρόπο στην καθημερινή τους ζωή ώστε να το εκμεταλλεύονται θετικά. Μία επιστημονική μελέτη λοιπόν για αυτό το θέμα πανευρωπαϊκή κατά το τέλος του καλοκαιριού ξεκίνησε και τα αποτελέσματα ίσως σε δύο χρόνια θα τα έχουμε στη διάθεσή μας. Και τότε θα έχουμε τη δεύτερη ανάγνωση που θα έχουμε ολοκληρώσει αυτού του νομοθετήματος εμείς. Δηλαδή αποφασίζουμε εμείς για ένα νομοθέτημα όπου λείπουν τα στοιχεία αυτά. Η βάση δεδομένων επιστημονική για το τι χρειάζονται οι καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε στο τι θέλουν οι καταναλωτές και στη συμπεριφορά τους και στις δικές τους συμπεριφορές για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, μία ε, βάση για την ετικετοποίηση που πρέπει να είναι εύληπτη και κατανοητή. Πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν οι καταναλωτές τι αναφέρεται από πλευρά συστατικών και ουσιών Ποιο ξέρει όμως πόσο περίπλοκα γραφήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σχεδιαστούν. Διότι υπάρχει και τελείω διαφορετική κατανόηση στα κράτη-μέλη ενδεχόμενα για τέτοια πράγματα. Υπάρχουν γραφήματα και γραφική απεικόνηση του ενός ή άλλου είδους, διαφορετικές βέβαια μεταξύ τους στα κράτη-μέλη, αλλά όχι στο, τη συνολική επικράτεια ενός κράτους από κάποιες αλυσίδες καταστημάτων ή εμπόρων έχουν αναρτηθεί και από κάποιους παραγωγούς περιφερειακά σε κάποιες χώρες. Όλα αυτά θα πρέπει ως, ως πρόσθετα στοιχεία να επιτρέπονται εθελοντικά πρόσθετη εθελούσια επισήμαση, ετικετοποίηση. Πρέπει να είναι εφικτή εφόσον η υποχρεωτική επισήμαση δεν επικαλύπτεται από αυτήν και δεν παρεκκλίνουν τα στοιχεία και δεν παραπλανούν από την επίσημη υποχρεωτική ετικετοποίηση διότι τα γραφικά συστήματα, τα γραφήματα από κράτο σε κράτο και οι απεικονίσει είναι πολύ διαφορετικέ από κράτο σε κράτο. Δεν πρέπει να υπερφορτώνουμε τι ετικέτε υπερβολικά με πληροφορίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την άποψη «Α, οι καταναλωτέ δεν διαβάζουν τι βρίσκεται στις ετικέτε, γι' αυτό πρέπει να του υποχρεώσουμε να τα διαβάζουν». Γι' αυτό θα πρέπει στην μπροστινή σελίδα τους της συσκευασίας, ε, στο προστιόφυλλο να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Να μην το κάνουμε όμω αυτό λέω εγώ και μάλιστα στην ε, πρόσθετη σελίδα όλες αυτές τις πληροφορίες δεν θα διαβάζονται από τους καταναλωτές. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά σε ποιο σημείο της ε, συσκευασίας θα εντάσσονται ποιες πληροφορίες κιόλα. ποιες πληροφορίες που θα εντάσσονται. Πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη σελίδα της συσκευασίας έξι υποχρεωτικές ενδείξεις. Ενέργεια, λίπη και κορεσμένα λίπη, ζάχαρη, άλας, αλάτι. Πρόκειται εδώ και είναι απόλυτα σαφές για μια αρνητική επισήμανση για το αλάτι και τη ζάχαρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτέ τι δύο συστατικέ ουσίε τροφίμων τι εντόπισε ω βλαπτικέ, λέει. Βλαπτικέ, για οποιουσδήποτε λόγου. Γιατί το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται αλάτι. Το θέμα είναι σε ποια ποσότητα. Γιατί διαφορετικά εκείνο το οποίο θεραπεύει γίνεται φαρμάκι. Το φάρμακο γίνεται φαρμάκι. Είναι παλιά παροιμία. Αυτή την ξέρουμε. Αλλά αρνητική επισήμανση λοιπόν των δύο αυτών ουσιών, αλατιού και ζάχαρη. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπερβαρύνουμε την, ε, ε, την σελίδα. Και μάλιστα έλεγα κάτω δεξιά στις συσκευασίες, στην ίδια ε, περιοχή πάντα, να αναφέρεται και το περιεχόμενο ενέργεια σε θερμίδες αυτού του τροφίμου. Και έτσι μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν, μια και οι συσκευασίες είναι διαφορετικές. Για να υπάρχει αυτή η συγκρισιμότητα μεταξύ των στοιχείων αυτών, προτείνω σε θερμίδες το ποσοστό ενέργειας στην προστινή σελίδα ανά 100 γραμμάρια του προϊόντος ή 100 χιλιοστόλιτρα, 100 μιλιλίτερ, να αναφέρεται το, ε, η θερμιδική ε, περιεκτικότητα. Στην προσελίδα και όχι ταυτόχρονα όμως όλες ε, οι ενδείξεις των μερίδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ή ανά 100 γραμμάρια ή 100 χιλιοστόλιτρα ή ανα μερίδα στην την σελίδα. Εγώ λέω όχι. Ανά 100 γραμμάρια, 100 χιλιοστόγραμμα, χιλιοστόλιτρα με συγχωρείτε για τη συγκρισιμότητα. Αν υπάρχει όμως μία μερίδα μόνο στη συσκευασία, επιπρόσθετα τότε μπορούμε και υποχρεωτικά μπορούμε να πούμε η ε, θερμιδική περιεκτικότητα να αναφέρεται στην προστινή σελίδα, να μπορεί ο καταναλωτής με μια ματιά να δει τι θα καταναλώσω ως θερμίδες ενεργειακά παίρνοντας αυτή τη μερίδα ή αυτό το ποτό σε μια μερίδα ή όταν φάω αυτό το περιεχόμενο της συσκευασίας ή το πιο για τα ποτά. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αλκοολούχα ποτά να εξαιρούνται. Θέλει όμως μεικτά ποτά, μείγματα ποτών με αλκοόλ να τα καλύπτει. Πρέπει όμως να είμαστε συνεπείς. Αν τα περισσότερα αλκοολούχα θα εξαιρούνται και όσον αφορά όλα τα αλκοολούχα θα εξαιρούνται, τότε ρυθμίζονται ξεχωριστά. Εδώ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το βρίσκω σωστό, μετά από πέντε χρόνια να συνταχθεί μια έκθεση αξιολόγησης και να ξανασκεφτούμε τότε αν θέλουμε τα αλκοολούχα ποτά να επισημένονται στην ετικετοποίηση ξεχωριστά. Εγώ πιστεύω ότι τα αλκοολούχα δεν πρέπει εδώ να καλύπτονται, επειδή το αλκοόλ, το ενόπνευμα δεν είναι είδος τροφίμου, είναι είδο γευστικό που αφορά τι γευστικές επιλογέ. Και μπορεί κανείς να διαβάσει βρίσκονται ήδη στις συσκευασίες ότι ουσιαστικά τις υποχρεωτικές ε, ενδείξεις ε, μέγεθος τύπου, ψηφίων τύπου τριών χιλιοστών πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ακούγεται μικρό αυτό, αλλά για τις πάρα πολλές ενδείξεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ήδη πολύ. Ήδη από το lobbying θα έχετε κάποια παραδείγματα τα οποία θα είδατε χειροπιαστά πόσο, σε τι εύρος γίνονται αυτές οι υποχρεωτικές ενδείξεις γραφικά. Αν θέλει λοιπόν στα τρία ε, ε, χιλιοστά να το κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να μεγεθυνθεί, να μεγεθυνθεί σημαντικά η συσκευασία του προϊόντος. Και αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Εμείς εργαζόμαστε κατά των σκουπιδιών, περιττών προϊόντων συσκευασίας. Δεν θα πρέπει λοιπόν εδώ όσον αφορά τη συσκευασία που δεν είναι περιεχόμενο να καλύψουμε τέτοιες περιττές ενδείξεις και γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά και το μέγεθος των συσκευασιών αυτό θα οδηγούσε αν μεγεθυνθούν αυτές να βάζουν και μεγαλύτερο περιεχόμενο μέσα η παραγωγή, πράγμα το οποίο θα ήταν και αντιπαραγωγικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί στη συνέχεια τις ε, ήδη ε, ενδείξεις για αλλεργογόνα προϊόντα να αναφέρονται. Τα έχουμε ήδη δει αυτά σε σχέση με τις στατικές ουσίες. Θέλει τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα να τα εντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον κανονισμό. Θα πρέπει να καλύπτονται δηλαδή και να ρυθμίζονται με αυτόν τον κανονισμό φρέσκα, νοπά. Φρέσκα και νοπά, λαχανικά, φρούτα. Πώ θέλετε αυτά να τα ετικετοποιήσετε. Δεν γίνεται. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν εξαιρέσει για προϊόντα που κατά τη χρονική στιγμή τη πώληση δεν είναι συσκευασμένα. Εντάξει, εγώ βλέπω εδώ τώρα να υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι ίσω ε, κάποιο μικρομεσαίο ξεχνά να προσαρμοστεί και να συμμορφωθεί σε αυτή τη ρύθμιση. Ή περνάνε μήνε μετά την έναρξη σε ισχύ αυτού του κανονισμού και δεν το κάνει αυτό. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια μη συσκευασμένα προϊόντα μέχρι τη στιγμή μιας εθνικής ρύθμισης να πρέπει να υλοποιούν όλε τι προποθέσει και όρου που αποφασίζουμε και εγκρίνουμε εμεί με αυτόν τον κανονισμό και κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο. Οι αλλεργογόνε ενδείξει όμω, πιστεύω ότι είναι εφικτό να, να χρησιμοποιούνται και για τα μη συσκευασμένα προϊόντα. Για αυτά τα μη συσκευασμένα, για παράδειγμα, γεύματα από εστιατόρια, κηλικία, όπως και εδώ στο εστιατόριό μας, η κηλικείο μας στην Ευρωβουλή. Τα αλλεργογόνα για τις ενδείξεις τους πρέπει να αναφέρονται με κάποια σηματάκια ή με κάποιο τρόπο που θα δίνει μια επισήμανση στον πελάτη ότι το προσωπικό πώλησης μπορεί να τους δώσει πληροφορίες ή μέσω φυλαδίων που μπορούν να είναι διαθέσιμα. Δεν χρειάζεται να το κρεμάμε αυτό το, φυλα, το φυλάδιο στα προϊόντα αυτά, αρκεί το φυλάδιο αυτό ε, ως ενημέρωση να είναι διαθέσιμο. Προτείνει λοιπόν και εθνικά συστήματα ρύθμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούν λοιπόν τα κράτη-μέλη να έχουν ξεχωριστά δικά του εθνικά συστήματα επισήμανση και ετικετοποίηση, που όμω δεν θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Κρούω κόδωνα κινδύνου και γι' αυτό, να μην το κάνουμε. Ακόμα και αν εθνικά συστήματα de jure βάσει νομοθεσία δεν, θα είναι, δεν θα είναι υποχρεωτικά, λόγω τη de facto εφαρμογή εκ των πραγμάτων συμμόρφωσης θα δημιουργείται μια διχοτόμηση της αγοράς, της ενιαίας εσωτερικής αγορά, ένα κατακαιρματισμό της και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σε διαφορετικές περιοχές ε, και περιφέρειες πολλούν τα προϊόντα τους. Θα είναι δύσκολο να ξέρει κανείς σε ποιο κράτο μέλο ισχύει ποια εθνική ιδιομορφία από πλευρά νομική ε, ε, υποχρέωση για την ετικετοποίηση και αναφορά στοιχείων. Θα ήταν ένα είδο υποκατακαιρματισμού πολυθρηματοποίηση ε, σε θράψματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Να μην το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, τα μη συσκευασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό και καθώς και εθνικές ε, ε, ρυθμίσεις για τα συστήματα αυτά να μην επιτρέπονται ακόμα και μη δεσμευτικά εθνικά συστήματα γιατί διαφορετικά θα είχαμε μια χαοτική, χαοτική χαόδη κατάσταση στην Ευρώπη. Δεν θέλω να επισέλθω σε κάθε λεπτομέρεια της έκθεσης. Σε κάποια μικρά ελάσσον σημασία, ίσον σημασία θέματα θέλω να αναφέρω. Θερμιδική ε, περιεκτικότητα στην πρώτη ε, σελίδα της συσκευασίας και ή και στην πίσω ε, σελίδα, πίσω όψη, με ένα κουτάκι που μπορεί να επαναλαμβάνει τα στοιχεία αυτά, όπου θα αναφέρονται οι συστατικές ουσίες. Αυτά τα κουτάκια που έχουμε, τα τετραγωνάκια που έχουμε, οι ορθογόνια που υπάρχουν και που εθελοντικά αναφέρονται τα στοιχεία αυτά, τώρα θα είναι υποχρεωτική ένδειξη αυτή. Και εγώ πιστεύω ότι μόνο σε χιλιοθερμίδες, κιλοκαλορί λέει η ε, ομιλήτρια. Ξέρω ότι και σε κιλοζούλ αναφέρονται, αλλά, αλλά κανένας ε, καταναλωτής δεν μπορεί με την έννοια κιλοζούλ να κάνει οτιδήποτε. Κατανοούν την έννοια θερμίδες ή χιλιοθερμίδες. Τώρα, την έννοια κιλοζούλ τη θεωρώ προβληματική. Για διαφορετικά πολλούς αριθμητικούς και αριθμούς και αντιστοιχίες θα έπρεπε να αναφέρουμε για να εξοικειωθεί ο, καταναλωτής. Τα αναγκαία ορθά στοιχεία επαρκούν. Οκτώ στοιχεία ενεργειακή περιεκτικότητα, δηλαδή θερμιδική αναφορά, όλα με βάση τα 100 γραμμάρια ή τα 100 χιλιοστόλιτρα. Επίσης, το λεύκομα, με συγχωρείτε, οι πρωτεΐνες. Ε, οι πρωτεΐνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να αναφέρονται. Όμως οι πρωτεΐνες είναι ένα από τα σημαντικότερα ε, στοιχεία στα τρόφιμα. Και έχουμε φυσικά και το θέμα της, ε, της τροφικής ανταπόκρισης για κάποιες ομάδες πληθυσμιακές είναι σημαντικό να μπορούν να έχουν υψηλή πρωτεϊνούχα τροφή που θα καταναλώνουν και γι' αυτό παρακαλώ να συμπεριληφθεί. Μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τι θα αναφέρουμε τα υδρογονούχα, τους υδατάνθρακες, με συγχωρείτε, ε, και μάλιστα και από ζάχαρη ή πώς. Προτείνω να το κάνουμε αυτό. Το επόμενο ερώτημα, τι θα κάνουμε με το αλάτι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το αλάτι. Δεν είναι πιο σωστό να αναφέρουμε το το νάτριο. Αλλά το αλάτι δεν είναι νάτριο. Δεν είναι όλα όσα περιέχει το αλάτι νάτριο. Υπάρχουν άλλες πηγές νάτριου στην ε, φύση και στη ζωή πέρα από το αλάτι. Ή θα πρέπει να αναφέρουμε αποκλειστικά μόνο το νάτριο, πράγμα το οποίο δεν θα κατανοούν οι καταναλωτές ούτως ή άλλως, ή θα αναφέρουμε στην επισήμαση νάτριο και ως υποσημείο, υποκατηγορία, από αλάτι ως πηγή Ίσως έτσι θα είναι πιο κατανοητά. Μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα με κατανοητό, εύληπτο τρόπο. Για τα τρία χιλιοστόμετρα, για τους, τα ψηφία της, ε, που θα τυπώνουν ε, αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει ακόμα τέτοιος ε, ορισμός, αλλά ένα κείμενο το οποίο είναι και πολύ μικρότερο από τρία χιλιοστόμετρα στα ψηφία του, πάλι εύκολα μπορεί να αναγνωστεί αν κάποιοι παράγοντες υλοποιούνται. Η αναγνωσιμότητα δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων, αλλά και από την αντίθεση των διαφορετικών χρωμάτων ε, που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία το, το είδο συσκευασία κτλ. Προτείνω με τις επιχειρήσεις να εκπονηθούν οι σωστές κατευθυντήριε γραμμές τι θα γίνεται με το μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκπροσώπους των παραγωγών τροφίμων πρέπει να καθορίσει ρεαλιστικό μέγεθος των ψηφίων, τυπογραφικών ψηφίων. Διότι πιστεύω ότι αναμερίδα, για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρεται η θερμιδική περιεκτικότητα πέρα από τις υποχρεωτικές ε, ενδείξεις που πρέπει να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, αλλά τι είναι μία μερίδα. Πώς μπορεί να καθορίσει κανείς ε, ή πόσο μεγάλο είναι ένα κουτάλι ε, του τσαγιού ε, πρέπει κανείς αυτά τα πράγματα να μπορεί με ρεαλιστικό τρόπο να τα ρυθμίζει, διότι διαφορετικά είναι παραπλανητικά. Είναι πολλές φορές ε, η περίπτωση που παραπλανούνται οι καταναλωτές με το μέγεθος μερίδων και τα λοιπά. Εγώ είμαι κατά της παραπλάνησης ως θέμα αρχής. Υποβάλλω πρόταση πώς ε, μπορούν σε σχέση με τα τρόφιμα, τα νητράτα και τα, αυτές οι συστατικές στοιχείες να καθορίζονται και μάλιστα θέματα που στην κοινή συζήτηση, στην δημόσια συζήτηση δεν είχαν προαχθεί. Τώρα έχουμε μεγάλη συζήτηση στην ε, Γερμανία και όσον αφορά την ε, χρήση αυτών των ουσιών, για παράδειγμα, Υπάρχουν τυριά που αποκαλούνται, τα αποκαλούμε τυριά χωρίς να είναι τυριά, διότι παράγονται από φυτικά λίπη. Αυτά στην πρόστια όψη πρέπει να αναφέρονται. Αν κάτι είναι απομίμηση τροφίμου, παράδειγμα, ή μια συστατική ουσία που αναμένει κανεί να την βρει σε ένα τρόφιμο, αντικαθίσταται ως, από ένα υποκατάστατο το οποίο είναι χαμηλότερη τιμή, είναι πιο φθηνό και το οποίο ο δεν ανέμενε να βρει μέσα σε αυτό το τρόφιμο που αγοράζει. Λοιπόν, αυτά είναι τα ουσιοδέστερα στοιχεία από πλευρά μου. Θα έχετε διαπιστώσει από όσα είπα ότι εγώ δεν είμαι υπέρ του συστήματο GDA ω υποχρεωτική σύστημα επισήμασης. Δεν το θεωρώ αξιόπιστο αρκετά και αρκετά αποδειγμένο. Είναι καλύτερα κατανοητό όσον αφορά την χρήση του ε, όμως σε σχέση με, την, ε, με τους σηματοδότες τους φωτεινούς που δεν είχαν επιστημονική τεκμηρίωση, αυτό έχει επιστημονική τεκμηρίωση. Εγώ όμως παρόλα αυτά δεν θέλω GDA επισήμαση. Ε, θα ήθελα, εθελοντικά ίσως, εθελούσια να μπορεί να γίνεται αυτό, αλλά με την αναφορά 2.000 θερμίδες την ημέρα ως ε, θερμιδικό περιεχόμενο και μέχρι τις 5.000 ε, θερμίδες ε, ή και παραπάνω να είχαμε μια, μια τέτοια αναφορά για αυτά τα στοιχεία, αυτό θα ήταν παραπλάνηση. Μια προσέγγιση όπως εμείς στη Γερμανία και σε άλλες χώρες έχουμε συζήτηση για αυτά. Μια χρωματική ε, επισήμανση με χρώματα των προϊόντων δεν είναι ευταία και επιθυμητή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα προϊόντα. Θα οδηγούσε στο ότι βασικά τρόφιμα κατά κανόνα να έχουν ένα σημαδάκι κόκκινο για παράδειγμα, έχει πολύ υπερβολικό λίπος ίσως το γάλα. Και έτσι θα το, το γερμανικό ψωμί σε σχέση με το νοτιοευρωπαϊκό λευκό άρτο έχει σχετικά πολύ αλάτι. Γιατί εδώ έχουμε το θέμα ε, της, ε, του πώς το ψήνουμε το ψωμί μας. Και όλα αυτά την ε, χρωματική επισήμανση με μόνο αυτά τα τρία χρώματα πράσινο, κόκκινο, κίτρινο δεν θα ήταν ευκταία. Και τώρα όσον αφορά την χρήση ουσιών, συστατικών ουσιών ε, σε σχέση με τα τρόφιμα, για παράδειγμα ένα τυρί το οποίο έχει παραθεί από ε, φυτικό λίπος ε, θα είχε καλύτερες τιμές όσον αφορά ε, τα φυτικά λίπη από ότι ένα πραγματικό τυρί. Τι θα λέγαμε εκεί, ότι μακροπρόθεσμα θα λέγαμε ότι συνιστούμε την κατανάλωση αυτού του ψεύτικου τυριού. Λοιπόν, φτάνω τώρα στο θέμα της, του χρονοδιαγράμματος παράταση της ε, διορίας ε, για τις τροπολογίες. Η 9η Δεκεμβρίου έχει σχεδόν φτάσει. Είναι τεράστιο χαρτοφυλάκιο αυτό βέβαια. Όμως πρέπει να πούμε ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στο τραπέζι μας εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν αλλάζεται κάτι στην έκθεσή μου. Αλλάζει κάτι από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα είχα αντίρρηση να μετατεθεί η διορία για την κατάθεση τροπολογιών αυτό θα μπορούσε να ήταν και αδιάφορο. Αν όμως θέσουμε υστερότερη χρονική στιγμή από την 9η Δεκεμβρίου, τότε δεν θα καταφέρουμε να έχουμε όλες τις γλώσσες ε, όσον αφορά τη συζήτηση το Γενάρη. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ή όχι, να το συζητήσουμε. Αν πούμε ότι εντάξει, να μην το συζητήσουμε το Γενάρη, να το συζητήσουμε το Μάρτιο στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Αυτό θα οδηγούσε πρώτη ανάγνωση όχι το Μάιο, αλλά μετά τις θερινές διακοπές. Να το σκεφτούμε αυτό σοβαρά λοιπόν αν το θέλουμε. Ευχαριστώ ευχαριστούμε συνάδελφε Ζόμερ για αυτή την εισαγωγή σε ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο θέμα και 212 τροπολογίες δικές σας. Δικές σας και μόνο. Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses ihre Bemerkungen machen. Περνάμε τώρα στη συζήτηση λοιπόν. Οι συντονιστές ε, στον πρώτο γύρο θα μπορέσουν να παρεύουν. Έχουμε πολλούς που ζήτησαν τον λόγο, σίγουρα. Και έχουμε χρόνο μέχρι τις 4.30. Τρία λεπτά ο καθένας θα ήταν το ευθετότερο. Εντάξει, Βήμε, λοιπόν, τρία λεπτά περίπου, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Τα τρία λεπτά για ένα τέτοιο θέμα είναι πάρα πολύ λίγα. Ευχαριστώ την συγκήτρια για το κειμενό της, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συμβολίτες και οι στόχοι είναι δύο. Πρώτα-πρώτα η απλούστευση της ηθικετοθεσίας, βελτίωση της ιστορικής αγοράς για το φαγητό και επίσης να έχουν οι καταναλωτές ε, τις αναγκαίες πληροφορίες για να κάνουν τις επιλογές τους. Πολλές φορές αυτά είναι συμπληρωματικά, πολλές φορές δεν είναι, άρα θα πρέπει κανείς να βρει την κατάλληλη ισορροπία. Καλή είναι η αφετηρία που έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνώ με κάποια θέματα και με άλλα όχι να σας πω σε τι συμφωνώ. Να μην είναι προσυσκευασμένα τα τρόφιμα, έχει δίκιο η συγγήτρια, ακριβώς όπως τώρα είναι η πρόταση, είναι σαν θα πρέπει για τα πάντα να υπάρχουν πληροφορίες ε, διατροφικές, όμως αυτό είναι δυσανάλογο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τα ίδια και για τα προσκευασμένα για όλα επίσης. Ε, ε, το έτοιμο για παραπάνω πληροφορίε, αφιτηρία θα πρέπει να είναι το να αναφέρονται τα αλλεργεγόνα. Τώρα, όσον αφορά ε, τι πληροφορίε, ανά 100 γραμμάρια, προσοχή. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι θα πρέπει να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει διαφορετικά προϊόντα και γι' αυτό καλύτερα να έχουμε ένα χιλιόλιτρο ε, την, ε, την αναφορά αυτών των διατροφικών στοιχείων. Και να είναι αναμερίδα όταν έχουμε προσκευασμένες μερίδες. Και να μην αντικαθιστά όμω την, την διατροφική αξία, η θρεπτική αξία ανά 100 γραμμάρια, αλλά να είναι πρόσθετο για τα νανοστοιχεία τώρα και την ετικετοθεσία της υγεία και για τα κατεψυγμένα. Καλή ιδέα. Θα κατεβάσω πάντως κάποιες τροπολογίες και τώρα όσον αφορά τη χώρα παραγωγής, τη χώρα προέλευσης. Θα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές από πού προέρχεται και τα τρία δύο καταναλωτών θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δική μας χώρα να λέει η ετικέτα τα γαλακτοκομικά, φρούτα, προκυπευτικά, πουλερικά να λένε από πού προέρχονται, πού γεννήθηκε το ζώο, πού μεγάλωσε, πού εσφάγει. Και το ίδιο να ισχύει, δηλαδή να αναφέρει την προέλευση και στα γεωργικά προϊόντα όσον αφορά τώρα το ενοπνευματόδη. Πάρα από τους τα λέει η συγκήτρια ότι θα βοηθούσε τους κατασκευαστές να ε, δίνουν το ενεργειακό περιεχόμενο. όμω ε, όμως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ε, τουλάχιστον στην ετικέτα αυτό το, το, το, ποστό σε αλκοόλ και το ίδιο για τους υδρογονάνθρακε. γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για του καταναλωτέ το, το, το, πόσο, πόσο αλκοόλ υπάρχει. Άρα αυτό να το λένε τώρα όσον αφορά την διατροφική αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εδώ πέρα κάποια ε, ερμηνευτική δήλωση. Λέει για τα GDAs. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω, η Ερνά που έγινε στο Βασίλειο λέει ότι ε, όταν ψωνίζει κανεί αυτό είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο δεν οδηγεί σε σύγχυση και θα χρειαστεί επομένως μια ετικέτα που να λέει GDS και να έχει σηματάκι σαν να ήταν φανάρι της τροχέας. Και να αναφέρεται το κάθε στοιχείο που έχει θρητική αξία και την ποσότητα. Ε, λίπη ε, και χωρισμένοι και αλάτι. ή να αναφέρεται μόνο η ενεργειακή αξία. Ούτως ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τις πιο υγιεινές επιλογές και να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους κατασκευαστές να μπορέσουν να προσαρμόσουν την παραγωγή τους ανάλογα. Αυτό ήδη γίνεται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, τα πρεσκευασία να υποχρεωτικά να αναφέρονται και άλλα θέματα υποχρεωτικά, όπως οι υδρογονάνθρακες, πρωτεΐνες κλπ. Τώρα το ευανάγνωστον. μέγεθος γραμμάτων, χρώμα στοιχείων και ε, το background σε σχέση με το χρώμα των γραμμάτων. Τι χρώμα θα έχει. Επομένως, να προβλέπονται κάποια ελάχιστα. Δεν αργό, δεν αργό, τελειώνω, τελειώνω. Αυτά τα, τεχνη, τα, τεχνικά, τα τεχνητά στοιχεία που θα περιέχονται θα πρέπει να αναφέρονται και για την εθνική νομοθεσία. Δεν θέλουμε να βάλουμε τον πύχη προς τα κάτω σε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Δεν θέλουμε να δεσμευόμαστε τον Βασίλειο από κάποιες ε, κατώς προδιαγραφές. Εναρμόνιση λέει για τις μερίδες η Κομισιόν. Μισό, μισό λεπτό λέει ο Μιλήτρη πόσο αυτό θα είναι εύληπτο σε σχέση με τις δαπάνες. Κοινό ε, σύμβολο να υπάρχει όσον αφορά την διατροφική αξία. Έχει κάνει η Κομισιόν κάποια μελέτη όσον αφορά τους δρογονάνθρακες και τους υδατάνθρακες και, το, και την αλκοόλη. Uh, Ευχαριστώ. Ε, θα πρέπει κάποιος να επικεντρωθεί σε κάποια από τα στοιχεία της έκθεσης. Ε, δεν γίνεται να τα μιλήσει, να τα πει όλα, γιατί αλλιώς δεν θα παρέμβουν όλοι. Δεν θα έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Ο κύριος Γκαμπάντη. Α, είναι δύσκολο να κανείς σωστά το όνομά μου. Γκερμπάντη. Ευχαριστώ την κυρία Σόμερ για την ε, σαφή της έκθεση. Ευχαριστώ για την, ε, το ζήλο που κατέβαλε για να ε, ξαναασχοληθεί με το θέμα μετά την πρώτη απόπειρα την, ε, της πρώτη ανάγνωσης. Οι φιλελεύθεροι σε γενικές γραμμές μπορούν να την υποστηρίξουν. Φυσικά έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η νομοθεσία είναι για την ενημέρωση των καταναλωτών. Δεν είναι για την προειδοποίηση ή το κρούσιμο του κόδωνα. Επομένως, η ενημέρωση θα πρέπει να είναι ως τον πιο αντικειμενική. Και, εν συνεχεία, ο κάθε καταναλωτής με ατομική επιλογή θα αγοράσει τα προϊόντα που του ταιριάζουν. Δεύτερον, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε έναν από τους λόγους για τον οποίο ε, γίνεται η απλούστευση αυτής της ε, νομοθεσίας το να κοιτάξουμε παράλληλα διάφορα νομοθετικά ε, κείμενα, αυτό είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση από πλευράς Κομισιόν. Έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Φτάνουμε πραγματικά στους ανθρώπους που θέλουμε να φτάσουμε με, με αυτού του είδους την επισήμανση. Ίσως αυτό το θέμα είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να διερευνηθεί τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την υγεία τους λόγω της πρόσληψης τροφίμων, ε, νομίζω ότι δεν ενημερώνονται σωστά με βάση τις σημερινές ε, ετικέτες. Κάποιες ερωτήσεις προς την εισηγήτρια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πιο σαφώς γιατί θέλετε να βάλετε και τις πρωτεΐνες στον κατάλογο και γιατί το, αντικαθιστάτε το αλάτι με τον άτριο. Αυτό αφορά τους ε, καταναλωτές, για τους καταναλωτές. <laughs> Είναι σαφές τι είναι αλάτι, αλλά δεν νομίζω ότι ξέρουν σαφώς οι καταναλωτές τι είναι το νάτριο. Το GTA τώρα. Νομίζω ότι είναι ένας απλός και σαφής τρόπος Επομένως, δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να διαγράψουμε την υποχρεωτική αναφορά του GDA. 100 ε, γραμμάρια ημερίδες. Προτιμώ τη λύση της κυρία Σόμερ. Αποφεύγει τον όχι και τόσο αντικειμενικό τρόπο που αντιμετωπίζουμε τώρα, ότι δηλαδή τελικά αποφασίζει η βιομηχανία τι είναι μερίδα, αλλά εσύ που το τρως δεν ξέρεις τι είναι. Ε, τα χρώματα του φαναριού δεν είμαι πολύ υπέρ των χρωμάτων αυτών. Είναι <clears throat> τόσο πλουστευτικά που δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Αφορά συγκεκριμένα τρόφιμα και τα στυλιτεύει και τα εστιάζει σε αυτά με τρόπο που δεν μ' αρέσει. Παραδείγματο χάρη το ψωμί και το γάλα μπορεί να πάρουν κόκκινη κάρτα, κόκκινο χρώμα. δεν νομίζω ότι είναι και τόσο το ψωμί και το γάλα. Μ' αρέσει ο τρόπος που ασχολείται η κυρία Σόμερ με τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Στην ε, προεκλογική ε, εκστρατεία το χρησιμοποίησαν αυτό το θέμα τα αντιευρωπαϊκά κόμματα. Δεν θέλουμε να συμπεριλάβουμε τα μη προσυσκευασμένα σε αυτό το νομοθέτημα τα εθνικά μέτρα, εθνικά σχήματα και προγράμματα θα μπορούσαν να, είναι, να γίνονται σε εθελοντική βάση από τον κλάδο. Δεν είναι υπέρ των εθελοντικών σχημάτων που προωθούν οι κυβερνήσει, γιατί αυτό είναι κατά τη εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι η εσωτερική αγορά θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα όλων μας. Πίτερ Υποστηρίζω και εγώ όλους τους προηγούμενους που χαιρέτησαν την εργασία της κυρία Σόμε. Ε, θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδίως όσες παράγουν μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ε, σε μικρές, από μικρές εταιρείες, ε, ΜΜΕ δηλαδή, την ίδια αντιμετώπιση με τις μεγάλες εταιρείες. Πώς θα μπορούσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις μεγάλες. Επίσης, το κιλοτζάρ δεν είναι επιτυχές, ας μην το χρησιμοποιήσουμε. για τους κωδικούς με χρώματα. Νομίζω ότι είναι παραπλανητική. Αν το γάλα για μωρά προσυσκευαστεί, θα πρέπει να βάλουμε ένα κόκκινο ε, χρώμα εκεί, λόγω του υψηλού περιεχομένου σε λίπος. Θα δίναμε λέει την εντύπωση ότι είναι ανθυγινό. Ε, διάφορες ε, ομάδες του πληθυσμού έχουν διαφορετικές ανάγκες ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Ε, επομένως, ας μην το προβούμε σε μια τέτοια αξιολόγηση. Επίσης, δεν νομίζω ότι την παιδική ταχυσαρκία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μέσω αυτού του συστήματος. Το βασικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει καν με τα τρόφιμα. Ξέρω ότι από επιστημονικές μελέτες τα τελευταία 15 χρόνια τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Ε, τα παιδιά ε, δεν τρώνε περισσότερη σοκολάτα, δεν ε, πίνουν περισσότερες λεμονάδες από 15 χρόνια πριν. Αυτό που αλλάζει είναι ότι κάθονται περισσότερες ώρες μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή στον υπολογιστή. Αλλάζουν τα πράγματα στην ηλεκτρονική σφαίρα. Και αυτό είναι ο λόγο που έχουμε μεγάλη αύξηση τη παιδική παχυσαρκία. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα μέχρι ενό σημείου. Δεν νομίζω ότι όλα ρυθμίζονται με την ετικέτα στα τρόφιμα. Και δεν νομίζω ότι θα επιλύσουμε και το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας έτσι. Ας είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα, τα σωστά παραδείγματα και να υποστηρίξουμε τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά δεν θα πρέπει να ξεγελιόμαστε ούτε εμείς, ούτε να ξεγελάμε άλλους, ότι με τη σωστή, με τη θαυμάσια ε, επισήμανση, ετικετοθεσία στα τρόφιμα, θα αντιμετωπίσουμε την παιδική παχυσαρκία. 185 Δεν ξέρω ποια νούμερα χρησιμοποιείτε ως ε, βάση. Λέει ο κύριος ε, Σλίτερ. Ε, δεν ξέρω αν έχει... Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ρενάτα Ζόμερ. Ε, θέλω να σας πω όμως ότι... Ε, την έλαβα προχθές στη Σουδική εκδοχή ε, και εξέτασα εντάχει τις 212 τροπολογίες. Ε, σας υπόσχομαι ότι δεν θα υποβάλω άλλες 212. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα νανοσωματίδια και το κείμενο 622-71. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, με τα οποία δεν συμφωνούμε παρόλα αυτά, κυρία Σόμερ. Ορισμένοι θεωρούν ότι η πιστοποίηση προέλευσης, ε, δηλαδή από πού προέρχονται τα στατικά του συγκεκριμένου εδόδημου, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, νομίζω ότι για το κρέας θα πρέπει να έχουμε ενισχυμένη ετικεταθεσία, να βλέπουμε το ζώο που γεννήθηκε, που ε, έχει ζήσει και που έχει σφαγεί. Και περιμένω μια πρόταση ε, της Κομισιόν για τους τροποποιημένους κανόνες για τη μεταφορά ζώων. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει νόημα να λέμε ότι γεννήθηκε στο Βέλγιο, ε, έζησε στην Ισπανία και σφαγιάστηκε στην Ολλανδία. Στην τροπολογία 106 αλλάξατε τον ορισμό της μικρής συσκευασία. Σημαντική είναι η αλλαγή που έγινε εδώ σε σχέση με, το με την αρχική πρόταση. Ε, πολλά, ε, πολλές συσκευασίες ε, ξερούνται από τις ε, απαιτήσει. Παραδείγματο χάρη για τα συστατικά. Από τα 10 τετραγωνικά εκατοστά πήγαμε στα 80 τετραγωνικά εκατοστά. Εγώ δεν είμαι κατά αυτή τη ιδέα 100%. Αλλά για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να, το έχουμε, να λάβουμε κάτι υπόψη μα. Αν κάτι προέρχεται από την περιοχή σου, θα μπορούσε να ρωτήσει ε, του βοηθού στο μαγαζί, το προσωπικό. Ε, σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεσαι ετικέτα. Αλλά όταν ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο, τότε ο καταναλωτή δεν έχει άλλο τρόπο να ενημερωθεί παρά μόνο την ετικέτα. Δεν μπορείτε να μειώσει τι απαιτήσει για τι ε, ετικέτε ε, παρά μόνο όταν βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη περιοχή ε, για την τοπική παραγωγή. Τώρα, για τα γλυκαντικά. Θα ήθελα πιο σαφείς κανόνες. Εγώ σε κάποια φάση νόμιζα ότι αγόραζα πραγματικό ε, χυμό πορτοκάλι, ενώ στην πραγματικότητα ε, ήταν γεμάτος από ζάχαρη. Μπύρα, κρασί και πνευματόδη. Μπορεί κάποιος να είναι αλλεργικός και σε αυτά, όπως μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο. Και αυτά είναι αλλεργιογόνες ουσίες. Ε, η μπύρα επίσης έχει πάρα πολλά οι Σουηδοί ε, γιατροί λένε ότι μπορεί κανείς να πιει κρασί, κρασί ε, ή να φάει σοκολάτα. Αλλά αν πίνει συστηματικά κρασί, ε, παίρνει πάρα πολλά καλωρί χωρίς να το γνωρίζει. Επίσης θα πρέπει να ε, επιχρεώνουμε να μπαίνουν πληροφορίες για το ποιοι ε, παραγωγοί χρησιμοποιούν φυσικές μεθόδους παραγωγής και ποιοι όχι. Τελειώνω, ε, τελειώνω ναι. Ε, στους πράσινους συζητήσαμε πάρα πολύ το θέμα των κωδικών με χρώματα, όπως ε, τα φανάρια της τροχέας. Νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος για να παίρνουμε πληροφορία ε, πολύ γρήγορα. Αν προσθεθεί όμως στις πληροφορίες ανά 100 γραμμάρια ή αν 100 μιλιλίτρ. Και για να αποφύγουμε τα γελία παραδείγματα που ακούσαμε για το γάλα σε σκόνη, ας πούμε. Ε, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να, αφορούν, να μόνο τα προσυσκευασμένα προϊόντα. σε ευχαριστώ. Σε μας λέμε τρία ποτήρια μπύρα είναι ένα κιλό ψωμί. Μπορεί κανείς να πει ότι με την μπύρα αντικαθιστά τρόφιμα. Είναι τρόφιμο. Για το κρέας ε, ο χαρακτηρισμός προέλευσης είναι απλούστερο. Για το φρούτο στα γιαούρτια είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Ή για το αμύγδαλα στις σοκολάτες όταν οι πρόσθετες, τα πρόσθετα υλικά προέρχονται πότε από τη μία χώρα, πότε από μια άλλη. Ε, τότε εντάξει, θα μπορούσε κανείς να το αναφέρει και αυτό. Κατή τα παρακαλώ. Yeah, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω στην κυρία Ζόμερ ότι το βρίσκω πολύ θαραλέο ότι έδωσε συνέχεια σε αυτό το θέμα, διότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία επί χρόνια εργαζόμαστε. Υπήρχαν τόσες πολλές τροπολογίες. Είναι θαραλέο, γενναίο το ότι έδωσε συνέχεια σε αυτό και το ανέλαβε. Ξέρει ότι διαφωνώ μαζί της. Σε κάποια σημεία συμφωνώ, σε άλλα βέβαια όχι. Λοιπόν, η δική μου πείρα ποια είναι. Όσον αφορά την τελευταία εξέταση αυτή της έκθεσης. Πολλές τροπολογίες απέρευσαν από το ότι σε αυτή την έκθεση ασκείται μεγάλη λομπιστική δραστηριότητα. Θέλω σε κάθε έναν που εργάζεται για αυτή την έκθεση να θυμόμαστε ότι πρόκειται εδώ για πληροφορίες για τους καταναλωτές και τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θέλω να επισημάνω ότι το λόμπι που αυτή τη στιγμή δρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απορριθμιστεί. 80% των λομπίστων είναι από τον τομέα αυτών και 5% των λομπίστων προέρχονται από τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών. Οι υπόλοιποι είναι των παραγωγών που πραγματικά δηλαδή να ενδιαφέρεται κάποιος για τους καταναλωτές. Πολύ λίγοι, 5%. Ελπίζω ότι θα εισακουστούν πολύ περισσότερο οι 5% από τους εκπροσώπους των βιομηχάνων, διότι εδώ έχουμε συμφέροντα καταναλωτών που πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα και κύρια. Αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, μίλησα με μια σειρά ενώσεων ε, καταναλωτών και συλλόγων και πολλοί από αυτούς δεν συμφωνούν. Δεν συμφωνούν το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη ότι δεν δηλαδή το εκτιμούν, λέει, οι καταναλωτές. Καθόλου. Υπάρχει μια σειρά χωρών όπου αυτό το σύστημα κωδικοποιημένο σε τρία χρώματα στα χρώματα των σηματοδοτών λειτουργεί και είναι πολύ θετική η ανταπόκριση των καταναλωτών. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν το βλέπω όπως η κυρία Ζόμερ. Δεν βλέπω την αρνητικό αυτό το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών στα τρία χρώματα. Είναι μια δυνατότητα ώστε στην πρόσθεα όψη της συσκευασίας να ενημερώνονται οι καταναλωτές. Μετά, πιστεύω μετά ότι μια ολόκληρη σειρά ουσιοδών στοιχείων όπως ζάχαρη, λίπη, αλάτι και θερμιδικό ε, περιεχόμενο πρέπει να αναφέρονται στη σελίδα αυτή, στην όψη αυτή. Και αν υπάρχει μύτος της Αριάδνης, οδηγός, Κάθε ένας γνωρίζει αν υπάρχει υπερβολική ζάχαρη ή υπερβολικό αλάτι σε κάποιο τρόφιμο ότι δεν είναι υγιεινό. Όμως οι καταναλωτές θα έχουν την ελευθερία επιλογής. Παρόλα αυτά να αγοράσουν για παράδειγμα και να καταναλώσουν μια ε, σοκολάτα. Αλλά με την ενημέρωση θα είναι πιο εξοικειωμένοι και ενημερωμένοι. Δεν πιστεύω ότι όλα πρέπει να εναρμονιστούν καθόλου. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν την δυνατότητα στη διακριτική τους ευχέρεια, στη διάθεσή τους κάποιες ε, αναφορές στην, οπίστια, στην ε, οπισθοσελίδα, στην οπίστια όψη της συσκευασία να αναφέρουν. Αυτό πρέπει να μπορούν να το κάνουν. Συμφωνώ όμω με την κυρία Ζώμερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα παραδοσιακά προϊόντα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να καλύπτονται. Πρέπει να μεριμνήσουμε η έννοια μικρομεσαίος επιχειρηματίας και μικρομεσαία επιχείρηση μέχρι 200 δηλαδή 50 συνεργάτες ή εργαζόμενους. Δεν, εν, δεν εννοώ αυτούς έτσι, μέχρι 250 εργαζόμενους, ενώ τους μικρομεσαίους, μικροφουρ, ε, τους μικροφούρνους, μικροατοπία, βιοτεχνικής παραγωγής και άλλα τέτοια εργαστήρια. Αυτά πρέπει να μπορούν να εξαιρούνται. Μετά με την κυρία Ζόμερ. Όσον αφορά ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων της Επιτροπής που διαγράφησαν, είμαι υπέρ των διαγραφών, διότι οι διαγραφές πολλές φορές απλουστεύουν τα πράγματα και έχουμε ένα μικρότερο όγκο πληροφοριών που πρέπει να ε, επεξεργαστούμε σύμφωνοι. Καμιά φορά όμως με τις πολλές διαγραφές χάνουμε την ουσία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ δεν θα συμφωνούσα να απολεστεί η ουσία. Αυτά γιατί διαφορετικά δεν θέλω να επισέθω σε λεπτομέρειες γιατί θα χρονοβορούσα, μακρηγορούσα. Πιστεύω λοιπόν ε, συνοπτικά ε, περιλήψει ότι πρέπει να προβληματιστούμε και να λάβουμε υπόψη ότι ο καταναλωτής θεωρεί με θετικό τρόπο αντιμετωπίζει τους σηματοδότες τα τρία χρώματα ε, ως κωδικοποιημένες αναφορές και δεν πρέπει να παραπλανούμαστε από λομπιίστες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του, των επιχειρήσεων του τομέα. Διότι δεν πρόκειται για αυτό, αλλά για την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Οι σκιώδεις εισηγητές ε, ήταν αυτοί, πέντε λεπτά είχαν στη διάθεσή τους. Τώρα έχουμε 13 που θέλουν να παρέμουν. Κλείνουμε τον κατάλογο και απευθύνω έκκληση μεταξύ δύο και τριών λεπτών ε, η παρεμβάση σας. Δεν χρειάζεται όλα να επαναληφθούν ε, σε παρατηρήσεις όσα έχει κανείς να πει. Μπορεί κανείς να είναι συντομότερος. Διαφορετικά μπορούν να συνταχθούν τροπολογίες. Ίσως και να διατυπώσετε ερωτήσεις προς την εισηγήτρια, αν γίνεται αυτό. Η κυρία Ντάγμα Ροτμπέρεντ παρακαλώ πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε αμέσως ευθύς εξ αρχής μετά την κυρία Λεωτά, Λομπίστες δουλεύουν πάντα για κάθε νομοθέτημα. Κάθε ένας πιστεύει ότι πολύ εξυπηρετεί όταν ε, τον αφορά κάποιο θέμα να εμπλέκεται. Εδώ και πολλά χρόνια όλοι μας ασχολούμαστε με την πολιτική για τους καταναλωτές. Αυτό πρέπει να είναι το μέρη, η μέρημνά μας, το μέλημά μας. Να υπογραμμίσουμε ότι αυτό εδώ είναι ένα νομοθέτημα που καλύπτει ένα κενό δεν έχει καμιά σχέση με οτιδήποτε άλλο. Δεν σχετίζεται αν είμαστε κατά της παχυσαρκίας, για παράδειγμα, ή για κάτι επιπρόσθετο. Κλείνουμε ένα κενό που υπάρχει, ένα χάσμα που μέχρι στιγμής για αυτή την ετικετοποίηση δεν υπήρχε κάποια πρόταση, κάποια ρύθμιση. Πρώτο και κύριο αυτό, αυτό χρειαζόμαστε το συνολικό πακέτο της επισήμασης των προϊόντων για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, ώστε να είναι ένα σύνολο εύληπτο. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Αυτό είναι η ευθύνη και ε, το καθήκον μας. Όταν το ξέρουμε αυτό είναι το επόμενο ερώτημα τι χρειάζονται οι καταναλωτές, τι θέλουν να γνωρίζουν. Θέλουν να γνωρίζουν ποιο ποσοστό τροφής και ποιε ουσίες εμπεριέχονται. Καλή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στρέφομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοιτάζω τους κυρίους εκπροσώπους που μπορούν βέβαια πολλά πράγματα να βελτιωθούν. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχεται ένα προϊόν. Στην εποχή των τρελών αγελάδων ήταν αυτονόητο το βόλιο κρέας να επισημαίνεται όσον αφορά την προέλευσή του. Γιατί να μην το κάνουμε και για άλλα. Είμαι υπέρ ένα κύριο τμήμα να το λάβουμε γι' αυτό, προσπάθεια δηλαδή καθορισμού προέλευσης και να κάνουμε να καταβάλουμε την προσπάθεια ώστε ο χαρακτηρισμός προέλευση για μια χώρα να λαμβάνεται υπόψη. Όταν για παράδειγμα καθορίζουμε τις ε, ε, ουσιώδεις ουσίες ε, και τα συστατικά όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το δούμε και το άλλο. Η συγγήτρια το διέγραψε αυτό ως πρόταση. Λυπούμε για αυτό που το διέγραψε την ιχνηλασιμότητα προέλευσης. Μετά, αναφορά πρωτεϊνούχων, πρωτεΐνης. Σε μια πρώτη προσπάθεια στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία είχα καταθέσει μια τροπολογία, τώρα την έχει κάνει δεκτή η συγγήτρια. Πιστεύω ότι είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία για τους ε, καταναλωτές. Ιχνοστοιχεία, στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη διατροφή και ασθενών. Νομίζω ότι και στο άρθρο 29 οπωσδήποτε και για τη χολυστερίνη πρέπει να αναφέρονται. Δύο στοιχεία είναι σημαντικά. Η διαφοροποίηση μεταξύ συσκευασμένων και μη συσκευασμένων προϊόντων. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί στην υπεραγορά, στο, ε, στο σούπερ μάρκετ πρέπει να αγοράζω ένα, μια μικρή ποσότητα σαλάτας όπου δεν αναφέρεται τίποτα και δεν υπάρχει συσκευασία. Λίγα βήματα παραπέρα υπάρχει συσκευασμένο από την εταιρεία φένιχ και όλα πρέπει να αναφέρονται ως συστατικά. Γιατί γίνεται το ένα και το άλλο όχι. Τουλάχιστον η, τα, αλλεργ, και για την ε, αναφορά τους και στα μη συσκευασμένα που πρέπει να αναφέρονται σε πολλά εστιατόρια είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Γιατί στο κηλικείο και στο εστιατόριο του κοινοβουλίου δεν γίνεται. Μετά, ε, γεύματα σε αεροπλάνα και αλλού μπορούν να εξαιρούνται. Όμως αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Σλούτερ, είναι 80 τετραγωνικά εκατοστά στο εμβαδόν τους. 80 τετραγωνικά εκατοστά, άμα το δει κανείς. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Θέλουμε να έχουμε τέτοια πράγματα όσον αφορά ε, την ε, συσκευασία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. πολλά έχουν υποθεί, κυρία Πρόεδρε. Ε, συγχαίρω την κυρία Ζόμερ που έκανε μια τεράστια δουλειά. Ο αριθμός βεβαίω των τροπολογιών είναι εξίσου σημαντικός. Ε, θα είμαι πολύ γρήγορη. Θέλω να αποφύγουμε, μια και ζητούμε την καλύτερη, την ενημέρωση για τον καναλωτή, να αποφύγουμε λοιπόν οτιδήποτε είναι κόκκινο φανάρι, πράσινο φανάρι ή πορτοκαλί φανάρι. Γιατί δεν είναι καλή ενημέρωση αυτή για μια ε, ισορροπημένη διατροφή η οποία εξασφαλίζεται ε, μέσα από μια πλειάδα τροφίμων. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να τα συνοψίσουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις πληροφορίες με χρώματα. Οι μελέτες δείχνουν ότι αυτό το σύστημα ε, δεν βοηθάει το καταναλωτή γιατί ο καταναλωτής θέλει μια ισορροπημένη διατροφή. Θέλουμε να πλουστεύσουμε την ετικετοθεσία, ούτως ώστε να είναι εύληπτη, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε την νομοθεσία για το μέγεθος των γραμμάτων. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Για κάποια προϊόντα, οι απαιτήσει ε, σε ό,τι αφορά το μέγεθος των ε, γραμμάτων δεν είναι ρεαλιστικές, όπως ε, τα μικρά και σεδάκια γιαουρτιού και τις μικρές συσκευασίε. Εκεί δεν μπορούμε να τα γράψουμε όλα, δεν γίνεται να τα γράψουμε όλα. Επομένως πρέπει να είμαστε απλώ ρεαλιστικοί. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να αναφέρει ενέργεια, οι πρωτεΐνες, τα γλυκίδια, οι ζάχαρες, τα λιπίδια ε, τα και κορεσμένα α, λίπη. Υπάρχει και το πρόβλημα του αλατιού ή νατρίου που θα πρέπει να αναφέρεται πίσω στην ε, ετικέτα. Μόνο... Λοιπόν, αλάτι ή νάτριο. Το αλάτι είναι συστατικό το νάτριο όμως είναι ε, στοιχείο. Ε, το αλάτι είναι βασικό στοιχείο της διατροφής, αλλά όχι το μόνο. Και άλλα στοιχεία, και άλλα συστατικά δίνουν ε, νάτριο, όπως υπάρχουν ας πούμε, στο, μέσα σε κάποια λαχανικά, μέσα σε κάποια κρέατα, σε κάποια αυγά κτλ. Ακόμη και στα νερά, στα μπουκάλια νερών. Με ανθρακικό. Επομένως προσοχή. Για την προέλευση των τροφίμων τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε την προέλευση των τροφίμων, γιατί ο καταναλωτής ε, όλο και περισσότερο ενδιαφέρεται για αυτή την πληροφορία. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε και εδώ. Αν αναζητήσουμε την προέλευση και μόνο των τροφίμων, θα μπορούσε να αναγκάσει τον καταναλωτή να αναζητήσει μόνο αυτή την πληροφορία και να ξεχάσει κάποιες άλλες πληροφορίες που θα ήταν πολύ πιο σημαντικές για αυτόν και που θα του επέτρεπαν, και τελειώνω έτσι, να κάνει μία πιο εγνωσμένη επιλογή. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Όλγα παρακαλώ. Ευχαριστώ προσπαθήσω να περιοριστώ στα τρία λεπτά. Δεν θα αναφερθώ σε όλα όσα προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα από τον Σιώδη εισηγητή μου προαναφέρθηκαν. Πράγματα, πράγματα που προσυπογράφω απόλυτα. Έχω κάθε σεβασμό για αυτό το οποίο επιτελεί ως έργο η κυρία Ζόμερ. Είναι πραγματικά Ηράκλειος άθλος και υπάρχουν πολύ λίγα σημεία όπου διαφωνώ και δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Είναι και λογικά και συνετά όσα έχει συντάξει από πλευράς προσέγγισης κάποιες, ε, ας το πω, κριτικές παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη σωστότερη κατεύθυνση να είχαν ακολουθήσει η πρότασή τους, διότι κάποια, κάποια σημεία υπάρχουν όπου διαρωτώμε πραγματικά. Κάποιος ο οποίος συντάσσει τέτοιες προτάσεις πραγματικά βρίσκεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την υλοποίηση τέτοιων προτάσεων. Ξέρει τι γίνεται. Θα περιοριστώ σε πολύ λίγα σημεία. Στην αρχή κάπως τρόμαξα ότι η προσέγγιση των GDAs διαγράφησαν. Στο τέλος όμως κατέληξα στο συμπέρασμα μετά από μεγάλο προβληματισμό και πολλές συζητήσεις που έκανα ότι ήταν σωστό ότι έγινε αυτό. Διότι αν κοιτάξετε στο σούπερ μάρκετ ε, στα ράφια έχω την εντύπωση ότι αυτή η προσέγγιση GDAs που είναι καλύτερη και πιο θεμελιωμένη από ότι οι φωτεινοί σηματοδότες ή αποτελούν αντικείμενο κατάχρηση από κάποιους παραγωγούς. Και εκπλήσωμε ότι μια ολόκληρη σειρά μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν κάνει τέτοιου είδου ε, λόμπι. Εδώ, για κοιτάξτε αυτό εδώ το προϊόν. Για την ένδειξη ποιες θερμίδε υπάρχουν με ενδιαφέρει ω 25 γραμμάρια λέει αυτής ε, της πλάκας ε, είναι 7% της ε, καθημερινής ανάγκης, ε, αν γυρίσω την άλλη πλευρά, 45 γραμμάρια διαβάζω. Πόσο λογική και συνεκτική είναι αυτή η πληροφορία που βρίσκεται σε αυτή την μπάρα σοκολάτας εδώ. Κοίταξα την προηγούμενη εβδομάδα και υπάρχουν πάμπολα τέτοια παραδείγματα. Έχω την υποψία, και να το πω αυτό πολύ προσεκτικά, ότι αυτή η μεγάλη υποστήριξη των GDAs των ε, ημερήσεων αυτών ποσοτήτων δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαφήμιση από τις ε, μεγάλες βιομηχανίες ε, και που εντάσσεται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Γι' αυτό ας επιστρέψουμε σε μια υποχρεωτική επισήμανση στις ετικέτες με δυνατότητα συγκρισιμότητας και σύγκρισης. Και όσον αφορά προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε κάνει, θα έλεγα πάντα πρέπει να είναι σαφές και να το συνειδητοποιούμε όλοι, το είπαν οι προλαλήσαντες, ότι με την επισήμαση τροφίμων και με τις ε, επισημάσεις στην ετικετοποίηση των τροφίμων, το πρόβλημα της κακής διατροφής δεν θα το επιλύσουμε. Δεν υπάρχει υγιές και μη υγιές τρόφιμο. Υπάρχει μόνο ισορροπημένη και μη ισορροπημένη συνήθεια όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες. Ούτε το ένα ή άλλο προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη υγιές. Αλλά όταν τρώει κανείς υπερβολικά από το ένα ή δεν τρώει καθόλου από ένα άλλο, τότε αυτό μπορεί να είναι βλαπτικό. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Μετά, όσον αφορά τους καταναλωτές, δεν πρέπει να τους χειραγωγούμε και να τους κυδεμονεύουμε και να επιβάλλουμε κάτι σε αυτούς ε, έτσι. Δεν μπορέσετε να τηρήσετε τα τρία λεπτά, πρέπει να σας ε, αναγκάσω να πειθαρχήσετε και να συμμορφωθείτε. Λυπούμε. Βάις Γκέρμπερ στη συνέχεια. Λυπούμε. Μόνο μία φράση να έλεγα. Έχουν ήδη περάσει και περίπου 10 δευτερόλεπτα του δικού μου χρόνου τώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου στου επένου προ την δική μα εισηγήτρια. Έκανε μια πολύ συνεκτική και λογική και πολύ σαφή έκθεση που μα υπέβαλε και που και εγώ 100% μπορώ να υποστηρίξω. Και αυτά που εγώ θέλω να συμπληρώσω είναι απλά συμπληρωματικές τροπολογίες που καμιά φορά μόνο σε συνδυασμό με τις προτάσεις τις δικές της μπορούν να λειτουργήσουν. Εκείνες που έχει εκείνη δεν θα τις ξανακαταθέσω εγώ, απλώς συμπληρωματικές τροπολογίες ε, έχω. Χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτό το οποίο έκανε όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Το βρίσκω καλό το ότι σε αυτό το σημείο εξαιρούνται αφορά αυτό ιδιαίτερα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφέρω μόνο τους, μικροφουρνα, τους μικροφούρνους ε, και ε, μικροπολία και μάλιστα με την, ε, φωτι... με την κωδικοποίηση των φωτεινών σηματοδοτών θα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα η νομοθεσία και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είμαι υπέρ της εθελούσιας, εθελοντικής επισήμασης και όπως το είπε σωστά ο Πρόεδρος πιο πριν σε σχέση με τους ε, ε, σοσιαλδημοκράτες, με τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι δύσκολο να δει κανείς από πού προέρχεται μια συστατική ουσία. Για τα νητράτα την πρόταση την βρίσκω καλή ώστε στην πρόσθετη σελίδα, πρόσθετη όψη να βλέπουμε ότι υπάρχει παρουσία νητράτων. Θα συμπληρώσω μόνο με έναν ορισμό και ένα παράτημα όπου τα παραδείγματα αυτά, οι περιπτώσεις αυτές θα αναφέρονται σαφώς. Δύο-τρία λόγια μόνο για τους σηματοδότες. Με τα επιχειρήματα που προαναφέρθηκαν είμαι και εγώ κατά των χρωμάτων των σηματοδοτών, διότι μπορεί να δημιουργηθεί και σύγχυση και λαθασμένη πληροφόρηση ή παραπλάνηση. Να νομίζει κανείς ότι πρόκειται για κάτι πολύ βλαπτικό. Ενώ εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε και να χτυπήσει συναγερμός. Γι' αυτό το σύστημα GDA το βρίσκω σωστό. Και εκείνοι που δεν το θέλουν και λένε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, το GDA είναι η μόνη εναλλακτική λύση στους σηματοδότες, δηλαδή ε, στο ε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Πρέπει μόνο να αποφύγουμε η βιομηχανία να ε, κάνει κατάχρηση του συστήματος GDA και να αναφέρεται σε συγκρισιμότητα ανά 100 γραμμάρια, 100 χιλιοστόλιτρα, η περιεκτικότητα, οι, και, οι θερμίδες κτλ. Έχουμε ένα, ένα πρότυπο πυλώνων ή αξώνων που θα μπορούσε να προταθεί. Ως πρόταση μόνο το αναφέρω και ως παράτημα θα το έβρισκα σωστό αν με σύστημα πυλώνων θα μπορούσε το σύστημα GDA να αναφέρεται στην επισήμανση και ε, μέσα σε αυτή την απεικόνηση να μπορεί αυτό να δίνεται στους καταναλωτές. σε ευχαριστώ. Βέσσερτ, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω καλύτερα με αυτό που οι κομματικοί συνάδελφοι από πλευράς της ομάδας μας δεν προανέφεραν. Ένα από τα πράγματα που η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ ήδη προανέφερε, δηλαδή το ότι κάποια τρόφιμα δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. Παράδειγμα, τρόφιμα, ε, μερίδες στο αεροπλάνο ή οι μερίδες που σερβίρονται σε νοσοκομεία. Και εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και αν δεν πληρώνει κανείς για τέτοιου είδους ε, διατροφή, έχει κανείς το δικαίωμα και θα πρέπει να έχει σίγουρα την δυνατότητα να πληροφορείται τι εμπεριέχεται σε αυτές τις μερίδες που του σερβίρουν. Σήμερα τι συμβαίνει. Διατάξεις υπάρχουν για τις ασπαρτίνες. Εμείς στο Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, είχαμε συνομοθετήσει και δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε αυτό το οποίο είχαμε κάνει στο παρελθόν. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μένα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει και επισήμανση και όσον αφορά τον Νικέλιο. Και επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει το θέμα. Εντάξει, και, και για τη ζάχαρη το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά και όσον αφορά τον Κέλιο. Είναι σημαντικό επιχειρήσεις και χώρες να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κάτι που θέλουν να καταναλώνουν οι καταναλωτές στη χώρα τους. Δεν πρέπει να είναι πρόβλημα αυτό αν κάποιες επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες των καταναλωτών και στις επιθυμίες τους, ίσως και πουλάνε περισσότερο από αυτό το προϊόν τους από ότι άλλοι που δεν συμμορφώνονται με, αυτές τις ε, επιθυμίες των καταναλωτών. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία της αγοράς και η ελεύθερη αγορά. Μετά, προέλευση, ε, προέλευση. Για το κρέα, παράδειγμα. Ακόμα και στη δική μου χώρα όμω δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει επισήμαση προέλευση. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί τα αλκοολούχα ποτά ξεχωριστά θα αντιμετωπίζονται. Αν είναι τρόφιμο ή όχι, είδο τροφίμου ή όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να εντάσσεται όμω μέσα σε αυτό το νομοθέτημα για τι ε, τροφέ, για τα τρόφιμα. Και όσον αφορά τώρα την, ε, ε, θρεπτική αξία, την θρεπτική αξία η ισοτιμία, ε, μέτρηση ε, της ε, θρεπτικής αξίας. Ανά 100 γραμμάρια, εντάξει, ή ανά 100 χιλιοστόλιτρα. Φοβούμαι ότι θα εξαφανιστούν όμως αυτές οι ενδείξεις αν συνέχεια φορτώνουμε και, και άλλες και καινούριε πληροφορίες στις ετικέτες. Τώρα, το να ξεκινάμε και να αναφέρουμε τα πάντα σε σχέση με 100 γραμμάρια ή 100 χιλιοστόλιτρα τα άλλα σε ποσοστώσεις ή σε περιεκτικότητα πρέπει να είναι συμπληρωματικά. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά και πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Αυτά τα οποία προανέφερα και είναι πιο σημαντικά. Τέλος, είναι σημαντικό τα ε, και κορεσμένα λύπη να αναφέρονται στην, ε, ε, στην ετικέτα. Και αυτά τώρα τα τρία χιλιοστόμετρα ή όχι για τα στοιχεία της εκτύπωσης δεν είναι το πιο σημαντικό αυτό, αλλά πάντα επαναλαμβάνεται σε επιχείρημα όταν μιλάει κανείς με τους πολίτες. Πρέπει να είναι ευανάγνωστα αυτά τα στοιχεία. Αυτό ζητούν οι πολίτες. Ευχαριστώ. Αντώνιο Παπαγνώβα, παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ως ιατρός θεωρώ ότι υπάρχει ένας βάσιμος λόγος για να θεπιστεί ένα τέτοιο νομοθέτημα και όχι μόνο για, την αθέμητη, τον ανταγωνισμό αλλά για λόγους δημόσιας υγείας διότι εάν όλα αυτά τα συστατικά τα ξέρει ο κόσμος είναι προειδοποίηση. Αποφύγουμε και το διαβήτη και την παχυσαρκία και, τα κυκλοφοριακά. Και όποτε παραπέμπουμε σε μελέτες που έχει κάνει η Φίλιπ Μόρις που λέει για το πόσο καλό κάνει το κάπνισμα στα δημόσια οικονομικά γιατί ο κόσμος πεθαίνει νέος. Πρόκειται και για τη στέγαση, για την κοινωνική πρόνοια, για το, σύστημα υγείας, για τη τεράστια ωφέλεια. Καμιά φορά επομένω το παρακάνει η βιομηχανία, μην ξεχνάτε. Άρα, όσο πιο πολλές πληροφορίε δώσουμε, καμιά φορά τους φέρνουμε μια σύγχυση. Άρα να λέμε μόνο για τα συστατικά τα οποία αφορούν την ημερήσια μία ε, λήψη. Και δεν είναι μόνο το νάτριο, είναι και η ζάχαρη και το αλάτι, όλα αυτά τα οποία έχουν σημασία. Να ξέρουν τις επιπτώσεις πάνω στην υγεία, εάν τα πούμε σωστά. Και αν κανείς είναι ειλικρινή, δεν χρειάζονται ούτε GDA, ούτε, ούτε φώτα της τροχέα, ούτε χρωματάκια, τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι το 10% των Ευρωπαίων είναι αναλφάβητοι. Και μόνο 10% έχουν κάποιο ανώτατο δίπλωμα. Όλοι οι υπόλοιποι απλώς δεν ξέρουν και πολλά για τα τρόφιμα. Μην ξεχνούμε επομένω ότι έχουμε αυτέ τι μελέτε και ε, καμία από τι τρει δεν αποδεικνύει το ότι δεν ωφελούν τα κίτρινα χρώματα πράσινα. Έχουμε όμως μια έκθεση από την Food Standards που λέει ότι τα GDS και τα χρώματα ε, μας οδηγούν σε, στην πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και άλλη μία έχουμε από Αυστραλέζικο Ερευνητικό Ίδρυμα που λέει ότι οι καταναλωτές πέντε φορές ευκολότερα μπορούν να βρουν τα υγιεινά προϊόντα όταν έχουμε τα χρωματάκια. Και επίσης, κατά τρίτον, έχουμε το δίκτυο για την πρόληψη των καρδιοπαθειών στην Ευρώπη. Και έχουν το πλέκτημα αυτά τα αισθήματα ότι μπορούν να μπουν σε όλα τα τρόφιμα και παντού. Άρα όλα αυτά μπορούμε να τα δώσουμε σε όλους και επομένως υπάρχει τεκμηρίωση. Άρα και τι είναι κατακλείδη όσον αφορά τα προφίλ, τα διατροφικά να τα χρησιμοποιεί ο κλάδος για τις διεθνείς τροφίμων για παιδιά. Υπάρχει νομοθεσία, ισχύει, δεν χρειάζεται την κατάσταση ισχύουσα νομοθεσία. Βιτόριο Πορι. Ευχαριστώ, Βιτόριο Πρόντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με τις ε, ονομασίες προέλευσης. Οι ονομασίες περιεχομένου θα πρέπει να έχουν γενικές πληροφορίες, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται μία ε, διατροφή ισορροπημένη, τουλάχιστον σε εβδομαδία βάση για τον καθένα μας. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τα διάφορα φανάρια της τροχέας, ειδικά με το κόκκινο χρώμα, γιατί σε αυτή την περίπτωση το αλάτι στις ε, σάλτσες παίρνει πάντα κόκκινο χρώμα. Φυσικά τις σάλτσες δεν τις τρώμε σκέτες, τις ε, βάζουμε συχνά πάνω σε λαχανικά. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια εξισορρόπηση της ε, διατροφής μας. Σάλτσες συν λαχανικά. Θα πρέπει να δίνουμε πληροφορίες και στα τρόφιμα τα οποία δεν είναι συσκευασμένα. Γιατί χάρη σε όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να υπάρχει μια ε, ισορροπημένη διατροφή. Κάτι που υπόθηκε πολλές φορές. Θα πρέπει να αναφέρουμε το περιεχόμενο σε ίνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ίνες για την πρόληψη διαφόρων ασθενειών του γαστεντερικού συστήματος. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε και κινδύνους για αλλεργίες. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Ε, υπάρχουν προβλήματα με το νοσοποιητικό σύστημα. Ε, οι αλλεργίες στις μέρες μας είναι όλο και πιο παρούσες, όλο και πιο σημαντικές. Επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν νόημα εάν ε, δίδεται στα πλαίσια μιας γενικότερης ενημέρωσης, ούτω ώστε η, η δίαιτα σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση να είναι ισορροπημένη. Ε, αλλιώς ε, οι πληροφορίες είναι εντελώς κατακαιρματισμένες και δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές. Δεν έχει νόημα και δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να φτάσουν σε μια υγιεινή διατροφή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αναεβδομάδα ή αναημέρα. Για ένδειξη. Αναημέρα νομίζω και όχι αναεβδομάδα, έτσι δεν είναι. Εγώ άκουσα ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς τι τρώει κανείς αναεβδομάδα ποσοστά οι, αυτές οι αναφορές είναι ημερήσιες αναφορές, έτσι, για ημερήσια κατανάλωση. Ε, για την εβδομαδιαία ε, διατροφή μιλούσα. Αυτή θα πρέπει να είναι, αυτή θα πρέπει να είναι ας πούμε η μονάδα μας, για, ε, η βάση μας. Αλλιώς δίνουμε κατακαιρματισμένες πληροφορίες, άχρηστες. Grazie. Corinne Lepage. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, λέει η κυρία Λιπάς. Έχουμε τρει στόχου οι οποίοι, οι οποίοι ακούστηκαν από πολλού συναδέλφου. Η υγεία και βεβαίω μπορούμε να τα λέμε όπω θέλουμε, αλλά το αλάτι, η ζάχαρη και τα λίπη δεν είναι οι μόνοι παράγοντε, αλλά είναι οι κύριοι παράγοντες ε, για την επιδημία παχυσαρκία στην Ευρώπη. Δεύτερον, η επιλογή του καταναλωτή. Να καταλαβαίνει τι επιλέγει να επιλέγει εγνωσμένα. Και τρίτον, η εμπιστοσύνη. Ε, Προηγουμένω κάποιο μίλησε στις, για τι τρελέ αγελάδε. Ε, εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στο προϊόν που αγοράζουμε. Εμπιστοσύνη στην προέλευσή του. Και να προσθέσω για κάτι άλλο. Το θέμα της προέλευσης σε σχέση με τον τόπο αγοράς ε, έχει μεγάλη σημασία και αυτό έχει σχέση και με τα περιβαλλοντικά θέματα και με το αποτύπωμα του διοξίου του άνθρακα. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφέρουμε την προέλευση. Νομίζω ότι ο φωτεινό σηματοδότη μπορεί να σα φαίνεται απλοϊκό, το είπαν κάποιοι, αλλά τουλάχιστον. Ε, μας λέει ε, λίγο, αρκετά ή πολύ. Αυτό σημαίνει τα τρία χρώματα. Δεν απαγορεύει τίποτα ο φωτεινός σηματοδότη. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους λιγότερο ενημερωμένους από εμά. Τρίτον, το είπαν και άλλοι, θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις. Δηλαδή, δόθηκε ένα παράδειγμα με την πλάκα σοκολάτας, ήταν σαφές. Ε, η μερίδα σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτή η μερίδα. Ας τα βάλουμε όλα ε, σε βάση 100 γραμμαρίων. Εν συνεχεία, θα πρέπει να δούμε τι είδους πληροφορίες θα δώσουμε για το αλάτι, ζάχαρη, πρωτεΐνες, ε, ίνες κτλ. Λαμβάνοντα υπόψη ότι όσο περισσότερο ε, βάζουμε στην ετικέτα, πιο δύσκολο είναι να την καταλάβουμε και να τη διαβάσουμε και να καταλάβουμε τα σημαντικά στοιχεία της. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του φωτεινού σηματοδότη είναι μια καλή προσέγγιση. Μια απλή και καλή προσέγγιση. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ε, πάμε να αποκτήσουμε μια κοινοτική νομοθεσία η οποία να είναι γενική, υποχρεωτική, ενιαία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διατροφική επισήμαση πραγματικά χρήσιμη. Και ε, δεν είναι τυχαίο ότι στόχος της έκθεσης Επιτροπής είναι να αντικαταστήσει αυτές τις επτά οδηγίες και τον ένα κανονισμό. Ε, επειδή άκουσα και για προθεσμίες ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο, μια εβδομάδα για τροπολογίες, θυμίζω ότι στην προηγούμενη προσπάθεια του 2008 ε, η πρώτη, η πρώτη μορφή της ε, πρώτης κανονισμού είχε συγκεντρώσει 1.332 τροπολογίες που δείχνει ότι οι 212 είναι απλώς μια καλή αρχή. Ακριβώς γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αναφέρει και η συγγήτρια, αλλά θέλουμε να προσθέσουμε. Ε, για, μας ε, είναι σημαντικό, για παράδειγμα, το ότι στις υποχρεωτικές πληροφορίες δεν μπορεί να εξαιρούνται τα αλκοολούχα, τα εινοπνευματόδη ποτά. Εδώ μπαίνει η επισήμανση σε άλλα ζητήματα. Άνθρωποι μπαίνουν φυλακοί σε κάποιες χώρες γιατί καπνίζουν κάναβη και εδώ δεν θα πρέπει να έχουμε μια υπόδειξη ότι μπορεί να, προωθ... να... να σμπρώξει κάποιον στον αλκοολισμό. Ε, επίσης, επιμέρους παρατηρήσεις κάνω, θα επιφυλαχθούμε και για ε, τροπολογίες. Ε, στην ε, τροπολογία 109 αναφέρεται για τα νανοσωματίδια, αλλά και πάλι παίζει το ρόλο του τροχονόμου. Ότι δηλαδή να προσθέσουμε τη λέξη νάνο. Χρειάζεται κάτι επιπλέον για αυτό το καινούριο και και εμφυλεγόμενη εξέλιξη στην, στον τομέα της διατροφής. Επίσης θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται μια ξεκάθαρη επισήμανση της χώρας προέλευσης. Χτες αναφέρθηκα πιο αναλυτικά σε αυτό. Ε, το συνδέουμε και με την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής. Με ενδιαφέρει ένα προϊόν ε, πέρα από το ότι μπορεί να έχει μια ποιότητα, να μην διανύει εκατοντάδες και χιλιάδες χιλιόμετρα για να έρθει ε, και έτσι να ε, επιδεινώνουμε και το φαινόμενο του θερμοκηπίου για τα ψάρια που ανήκουν σε πληθυσμού που απειλούνται θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στην ε, συσκευασία επίση, όπω ε, για τον τόνο συζητάγαμε. Οι γλυκαντικέ ουσίε θα πρέπει να αναγράφονται επίση ξεκάθαρα. Κάτι ακόμη. Ο όρο vegetarian δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροφές που περιλαμβάνουν υπολείμματα ζωικών ε, προϊόντων. θα ήθελα να πω ότι ε, είναι σημαντικό το ότι η συγκήτρια αναφέρει ότι η πρόταση κανονισμού έγινε χωρίς ε, τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε ε, πόση έκταση έχει. Πάντως θα πρέπει να τονίσω ότι για μας αν δεν υπάρχει μια απλή σήμανση όπως έχει προταθεί και από τον Γκάρτ Σλίτερ ε, από τους πράσινους για το, που να μοιάζει με, την, ε, με το φωτεινό σηματοδότη, τότε θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι το γεγονός το μέγεθο των γραμμάτων και ο όγκο των πληροφοριών δεν πρέπει να την πληρώσουν σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν πρακτικά αναλφάβητοι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλέ γλώσσε, υπάρχουν μετανάστε και θυμίζω, κλείνω, κλείνω, θυμίζω ότι υπάρχουν χώρες που αναβάθμισαν τις σκυλοτροφές okay. ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνταν από φτωχούς ανθρώπους. Χρειαζόμαστε σήμανση πιο απλή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φέστα Κλάς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την έκθεση Ζόμερ την βρίσκω καλή και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ζόμερ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ζήτησα όμω τον λόγο όταν άκουσα κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν στη συζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πράγμα πρέπει να έχουμε υπόψη μα. Μια ετικέτα δεν μπορεί να είναι εγχειρίδιο για υγιεινή διατροφή. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας, εντάξει. Και πρέπει να απόσχουμε από τέτοιου είδου φιλοδοξίε. Πρέπει να διαφοροποιούμε μεταξύ σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και επιπρόσθετων πληροφοριών που πρέπει να είναι εθελοντικού χαρακτήρα. Αυτές οι ελεύθερες πληροφορίες μπορεί κανείς και ως προτέρημα ανταγωνισμού, πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό να χρησιμοποιούνται από εκείνον που τις παρέχει. Όταν αγοράζει ε, ε, δεν αγοράζει ένα προϊόν όπου δεν αναφέρεται η προέλευση κάποιων ουσιών ή στοιχείων, ε, τότε λοιπόν προτιμά κάποιο άλλο το οποίο αναφέρει την προέλευση και αυτό είναι στοιχείο που ευνοεί τον ανταγωνισμό υπέρ του άλλου προϊόντος. Τώρα, όσον αφορά και τις θερμίδες, όπου πιστεύω ότι δεν χρειάζεται η αναφορά κιλοζούλ, δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν ως έννοια, ως στοιχείο αναφοράς, ας μην το χρησιμοποιούμε λοιπόν. Αλκοολούχα ποτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ειδικά εξειδικευμένους κανονισμούς, οδηγίες για υνοπνευματόδηποτα ποτά. Για το κρασί υπάρχει ειδική οδηγία ετικετοποίησης. Δεν είναι ότι δεν ετικετοποιούνται τα κρασιά στις φιάλες τους, όχι. Αλλά εδώ, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει μετά από πέντε χρόνια θα υπάρξει εκ νέου προβληματισμός, έχει κάποιο λόγο γι' αυτό, ώστε εμείς εδώ να μην χρειάζεται να αντιερχόμαστε σε σύγκρουση για αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν θα γίνει. Ευχαριστώ την Ρενάτε Ζόμερ για το ότι έχει συμπεριλάβει στην τροπολογία της ε, τα νητράτα, της νητρώδεις ουσίες. Ίσως θα πρέπει με σαφέστερο τρόπο να αναφερόμαστε εκεί όπου υπάρχει νητράτο, νητρώδης ουσία να αναφέρεται αυτό για την αρχή προέλευση Μπορεί να είναι μια εξαιρετική εθελοντική πρόσθετη πληροφορία, αλλά μόνο για το αρχικό ουσιώδες προϊόν ω τρόφιμο μπορεί να ισχύει, όχι για κάθε ουσία. Όταν έχουμε ένα προμαγειρευμένο προϊόν έτοιμο, πώς θα αναφέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, με βάση τον εθελοντικό χαρακτήρα αυτής της ρύθμισης για τον ανταγωνισμό θα ήταν μια καλή ε, ιδέα, θα ήταν θετικό ως πρωτοβουλία στον ανταγωνισμό να χρησιμοποιούν αυτές τι αναφορές προς όφελός τους εκείνοι οι οποίοι θα το κάνουν. Ευχαριστώ. Μπερλάτο παρακαλώ. You don't vote. Okay. Then, uh... Όχι, εντάξει. Esther Lange, παρακαλώ. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag eh, drie... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω. Πρώτον, σηματοδότες. Ο συνάδελφος από τους uh, σοσιαλδημοκράτες και άλλοι κάνουν σαν οι σηματοδότες να ήταν το μέσο για την καταπολέμηση λέει ή για την, τον αγώνα του φτωχού καταναλωτή κατά των μεγάλων λέει επιχειρήσεων και των λόμπι. Όμως ε, στην πρακτική εφαρμογή τι γίνεται και πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά να μην γίνουν παχύσαρκα διότι Διαφορετικά θα υπήρχε για παράδειγμα πράσινο σε κάποιο προϊόντα και μετά να, αφήνουμε, να πίνουν τα παιδιά κοκακόλα και να παχαίνουν και να αφήνουν το γάλα και τον ε, ε χυμό μήλων στο ψυγείο και να μην τον πίνουν. Ε, λοιπόν, γονείς που φοβούνται τα παιδιά τους να μην γίνουν παχύσαρκα εκείνοι είναι που πολλές φορές ε, αγοράζουν τέτοια προϊόντα, καταναλώνουν τα παιδιά Coca-Cola και δεν τρέφονται, δεν ε, διατρέφονται σωστά. Λοιπόν, δεν συσχετίζονται όλα αυτά με, τον, με, με το φταίξιμο των σηματοδοτών. Μετά, για τα μη συσκευασμένα και, προς και ε, συσκευασμένα που πρέπει να διαφοροποιούμε, δηλαδή για την χρήση κάποιων στοιχείων για τα προσυσκευασμένα και όχι για τα μη συσκευασμένα εξαρτάται από τον ορισμό. Είχα απασχοληθεί και σε κρεοπολείο παλαιότερα ή τι κάνει και κάποιος ο οποίος έχει, ε, είναι αρτοπόλης και κάποιος ο οποίος για παράδειγμα κόβει ψωμί, τα βάζει σε, το βάζει σε μία σακούλα και το πουλάει. Τι είναι, θεωρείται αυτό το προϊόν ε, ε, βιοτεχνικό προϊόν, θεωρείται προσυσκευασμένο ή όχι. Για μένα δεν είναι προσυσκευασμένο και πρέπει ξεχωριστά να αντιμετωπιστεί. Η κυρία Ροτ Βέρεν κάπως οργισμένα αντέδρασε, όμως έδωσε ένα καλό παράδειγμα από το Βερολίνο με εκείνη την πατατοσαλάτα που αναφέρθηκε. Λοιπόν, βλέποντας αυτό τώρα για μη προσυσκευασμένα τέτοια προϊόντα, για τα χιλικία, εστιατόρια, θερμιδική περιεκτικότητα κτλ. Αν θέλετε τα πάντα μπορούμε να απαριθμίσουμε και να αναφέρουμε. Εξαρτάται όμως αν αυτό θα είναι αποτελεσματικό ή όχι. Εμείς, εγώ είμαι από την Ολλανδία, δεν έχουμε τόσο μακρά παράδοση γαστρονομική όσο άλλες χώρες. Μέσω των βαθμών Μισλά που παίρνουν κάποια εστιατόρια έχουμε βελτιωθεί. Αλλά στη Λιόν και στη Γαλλία είδα ότι είναι υποχρεωτική αναφορά των θερμίδων. Τι γίνεται, λέει ο μάγειρα. Ξέρετε, αν κάθε φορά, για κάθε μερίδα πρέπει να κάνω υπολογισμό πόσε θερμίδε εμπεριέχει, δηλαδή και μάλιστα με εξαψήφια αναφορά μετά την υποδιαστολή χ ψηφία πιο πριν και μετά την υποδιαστολή άλλα να ακολουθούν, τότε έχουμε μια κατάσταση που υπονομεύει την γαστρονομική μας παράδοση. Δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Και έχουμε και τους ψηφοφόρους για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι. Όχι, δεν θέλουμε οι πολίτες μας να επιβαρυνθούν. Θέλουμε να έχουμε ε, τέτοια δημιουργικότητα στα εστιατόρια. ο Κρίστοφ παρακαλώ τελευταίο. Ευχαριστώ. Να μην να μην επαναλαβώ ότι προελέχθη, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι για τους καταναλωτές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπεραπλουστεύουμε, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν είναι ακριβή τα αναγραφόμενα. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κάτι ως, όπως ένα ε, τρόφιμο κακό ή επικίνδυνο. Άρα, να μην έχουμε ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί την εντύπωση ότι ένα τρόφιμο είναι κακό ή επικίνδυνο. Βεβαίω θα πρέπει να έχουμε ποικιλή στη τροφή μα, δεν πρέπει να τρώμε υπερβολικά και θα πρέπει να ασκούμεθα. Βέβαια δεν μπορούμε να τα λύσουμε με αυτή την οδηγία. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τον εαυτό του. Άρα μην αρχίσουμε να συμπεριφέρονται προς τον κόσμο σαν να πρόκειται περί λυθείων, γιατί τότε θα γίνουν οι λύθοι. Άρα με αυτή την οδηγία δεν θα πρέπει να δημιουργούμε μία πλαστή αίσθηση ασφάλειας. Δηλαδή θα πρέπει να κάτσουν να διαβάσουν τη λέει συσκευασία για να γίνουν υπεύθυνοι. Φυσικά και θα πρέπει κανείς να, να, να έχει ποικιλία διατροφής. Δεν θα πρέπει να τρώει πάρα πολύ και θα πρέπει να ασκείται. Ξέρω ότι οι πολιτικοί θέλουν να τα πάντα με κανονισμούς και με οδηγίες. Όμως, ε, να φτιάξετε ένα απλό μήνυμα, όχι δεν γίνεται αυτό, ξεχάστε το. Yeah. Σε ευχαριστώ. Ζωντανή και με πολλές, ε, θα έλεγα, συγκρόμενες απόψεις ε, συζήτηση. Θα δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν λάβει τον λόγο η συγγήτρια. Εσείς, κύριε Διευθυντά, για αυτό τον τομέα έχετε τον λόγο από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σας εκπλήξω αν σας πω ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για να πάρουμε στεναρές αποφάσεις, γιατί ο πρόεδρος Μπαρόζο μόλις ε, έχει διορίσει το νέο Σώμα των Επιτρόπων και οι νέοι επίτροποι θα έρθουν σε λίγες εβδομάδες, τον Ιανουάριο σίγουρα, ενώπιον του Κοινοβουλίου για τις ακροάσεις τους. Και εκεί θα πάρουν θέση για τα θέματά τους. Επομένως είναι δύσκολο σήμερα εγώ να σας απαντήσω έτσι πολύ λεπτομερώς σε όλες τις ερωτήσεις αλλά παρόλα αυτά μπορώ να κάνω κάποια σχόλια. Δεν θα σε εκπλήξει επίση το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν συμφωνεί με την ανάλυση της κυρίας Ζόμες για τη δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς. Δεν ε, συμφωνούμε και δεν συμμεριζόμαστε όλες τις προτάσεις της. Αντίθετα, πολλοί από εσά ε, ανέφεραν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την προέλευση ιδίω των προϊόντων. Πολλοί μίλησαν, όπως η κυρία Βίλμοντ, ο Σλίτερ, ε, η Ροτ Μπέρεντ, ε, η κυρία Λεπάζ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ε, θεωρούν ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν, δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη. Σε αυτό το κείμενο θέλαμε να λάβουμε υπόψη όλα όσα προϋπήρχαν ήδη, γιατί είναι ένα περίπλοκο θέμα, ένα δύσκολο θέμα και πάνω απ' όλα είμαστε προσεκτικοί και θα ακούσουμε οποιαδήποτε ιδέα, προσανατολισμό θέλετε να μας υποδείξετε. Η εγγραφή των συστατικών ε, στην εμπρόσθια, στο εμπρόσθιο τμήμα της ε, συσκευασίας. Θα πρέπει να μειώσουμε σε ένα τα ψηφία, θα πρέπει να έχουμε έξι ψηφία. Είναι δύσκολη η συζήτηση. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να βάλουμε αυτά τα έξι συγγνώμη, ε, στοιχεία. έξι στατικά, έξι στατικά στο τμήμα της ετικέτας, όχι ψηφία, συστατικά. Αλλά και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και ευχαριστώ την κυρία Γιωτέρα που με υποστήριξε για το μέγεθος των γραμμάτων. Το ανέφεραν πολλοί βουλευτέ αυτό το θέμα. Η κυρία Γκοστέτ ε, το ανέφερε για τα γιαούρτια στις μικρές συσκευασίε που πουλούνται. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε παρεκκλήσεις, ειδικά ε, για τα μικρά ας πούμε, τετραγωνίδια ε, βούτυρο που τρώμε στο, αεροπλάνο. Δεν μπορούμε ε, σε ένα μικρό τέτοιο κουτάκι, δύο επί 3 σαντιμέτρη να βάλουμε όλες τις πληροφορίες. Κάτι άλλο που είπαν η κυρία Κλάση, η κυρία Βάιτσμπεργκερ, είναι τα προϊόντα, τα ψευδεπίγραφα, οι απομιμήσεις. Εδώ σίγουρα θα πρέπει να νομοθετήσουμε για αυτά τα τυριά που γίνονται με φυτικά λύπη κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ τον καταναλωτή και του προκαλεί δυσκολία. Κάποια άλλα στοιχεία που έχουν ακουστεί. Ε, δεν θα θέσουμε σε αντιπαράθεση το GDA με το φωτεινό ε, σηματοδότη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το GDR, GDA συγγνώμη, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Δεν χρειάζεται να είναι μπροστά στην συσκευασία, μπορεί να είναι από πίσω. Αλλά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να εκτιμήσει την ποσότητα του προϊόντος σε σχέση με την ημερήσια πρόσληψή του για να δει αν απορροφά 5%, 10% ή 50% ε, καλωρία, ας πούμε, ή αλάτι, οτιδήποτε. Τώρα, ο φωτεινός σηματοδότης ε, είναι τμήμα των εθνικών σχημάτων, ε, των εθνικών προγραμμάτων που είναι εθελοντικά και δεν επιβάλλονται σε κοινοτικό επίπεδο. Πολλοί από εσά ε, μίλησαν για το πρόβλημα των ινών. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία των ε, ινών ε, για μια ισορροπημένη διατροφή και για μια καλή πέψη. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφέροντας αυτά που είπε η κυρία Ροτ Πέρεντ και η κυρία Λεπάζο για το νόημα αυτής της πρότασης το οποίο θα συνοψίσω ως εξής. Εμείς θέλαμε να έχουμε μια απλή, να υπάρχει μια απλή ετικετοθεσία, ευανάγνωστη, ε, τίμια και συγκρίσιμη. Για να καταπολεμηθούν διάφορες αρρώστιες, θέλουμε μια τέτοια ετικετοθεσία, αλλά κυρίως για να μπορεί να επιλέγει ο καταναλωτής. Φυσικά, δεν θα ρυθμίσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας των παιδιών με, μια τέτοια ετικέτα. Θα πρέπει να τα εμποδίζουμε να τρώνε α, αλατισμένους ξηρούς καρπούς, ε, θα πρέπει να τα εμποδίζουμε να βλέπουν συνέχεια τηλεόραση και θα πρέπει να τα οθούμε να τρέχουν. Για πολλούς καταναλωτές, είτε αλλεργικοί είναι, είτε όχι, είτε χρειάζονται ειδική διατροφή, είτε όχι είτε είναι πολύ δραστήριοι είτε κάνουν καθιστική ζωή, πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που προτείνουμε θα τους επιτρέψουν να κάνουν μια λελογισμένη επιλογή. Φυσικά χρειάζεται και παιδεία για κάτι τέτοιο. Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω το, τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους οποίους, εναντίον των οποίων βάλατε είναι δύο οι κυρίες αυτές οι οποίες δούλεψαν επί χρόνια για αυτό το θέμα. Δεν, μην φανταστείτε καμία στρατιά ευρωκρατών. Τις υποστηρίζω θερμά γιατί δούλεψαν με επαγγελματικότητα, με σοβαρότητα. Έγινε και μια μελέτη αντικτύπου, έγιναν διαβουλεύσεις πολύ έντονες ε, για όλους, με όλους τους ενδιαφερόμενους, τον κλάδο, το εμπόριο, τους καταναλωτές. Φυσικά ο καθένας έχει τελείως διαφορετικές και τελείως ε, δικές του θέσεις. Αλλά όλοι έχουν δώσει την άποψή τους στα πλαίσια της διαβούλευσης και πιστεύω ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν υπερβολικές, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πουλέ. Το ακούσαμε αυτό που αναφέρατε και όταν θα έχουμε τον νέο επίτροπο που θα προσέλθει για την ακρόαση και μπορούμε να διατυπώσουμε ερωτήσεις θα το κάνουμε. Κυρία Ζόμερ, θέλετε να αντιδράσετε στις παρατηρήσεις που ακούσατε. Τις επιθέσεις μου κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν τις αποσύρω. Δεν θέλω να επιτεθώ προσωπικά εναντίον σε κανένα. Όμως θα έπρεπε να έχει βασική στελέχη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε ένα ρεαλιστικό σχέδιο να έχει υποβάλει. Το σχέδιο το οποίο υπέβαλε δεν ήταν ρεαλιστικό. Και όταν λέει ότι από οι γνώμες εξωτερικών επαϊόντων δεν ήταν αναγκαίες, τότε διαρωτώ με πώς θεωρεί τον εαυτό της αυτοικανότατο για όλα τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς βοήθεια από οι Δήμονε. Θα έπρεπε και εξωτερικούς ε, πραγματογνώμονες να έχει χρησιμοποιήσει. Τώρα, δεν μπορώ να επιστρέφω σε όλες τις ερωτήσεις. Είμαι πρόθυμη να έχω προσωπική διμερή επαφή με όλους ε, όσους ε, έχουν κάποια θέματα. Όμως κάποια θέματα αρχής, πρώτον προέλευση πρέπει να αποσαφινιστούν εκτός από το κρέας και για τα συστατικές ουσίες τροφίμων, ουσιαστικές ε, συστατικές ουσίες τροφίμων. Αγαπητοί φίλοι, αυτό δεν είναι εφικτό τεχνικά. Αν έχουμε, την, έχουμε ένα ε, κέτσαπ προϊόν, ε, μπορούμε να έχουμε τομάτες από πάσης φύσεως ε, προέλευση, από κάθε χώρα του μεγαλοδύναμου. Και όσον αφορά τις άλλες ουσίες και τα, τις ζωοτροφές, παγκόσμια αγοράζονται αυτές οι πρώτες ύλες και το στοιχείο της τιμής, ε, της ευθυνής τιμής διαδραματίζει τον ρόλο του σε τέτοιες αγορές. Πώς μπορεί και όταν αγοράζουν ημερήσια κάθε μέρα διαφορετικές παρτίδες προϊόντων Πώς μπορεί για το τελικό προϊόν να είναι ηχνηλάσιμο από πού προέρχεται η ντομάτα ή κάτι άλλο. Εφικτό δεν είναι λοιπόν. Τώρα για το βόλιο κρέας έχει ρυθμιστεί, υπάρχει αυτή η επισήμαση από την εποχή των τρελών αγελάδων. Το υπόλοιπο κρέας. Ε, εδώ είχα, είχα υποβάλει μια πρόταση για στενότερη επισήμαση, την απέσυρα. Μου είπαν οι, ε, όσοι ασχολούν με την προστασία των ζώων ότι ο καταναλωτής δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει λέει στη συνέχεια κατά πόσον μεταφέρθηκε το ζωντανό ζώο σε σφαγείο για να σφαγεί, πράγμα το οποίο και αυτό θα ήταν σημαντικό στοιχείο. Εγώ θέλω να ξέρω πού ζούσε το ε, ζώο αυτό πριν σφαγεί και αυτό ίσως θα ήταν υπερβολική πληροφορία. GDA τώρα, Gross Daily Allowances, δεν είμαι υπέρ τη υποχρεωτικής ε, επισήμανσης. Και αυτό το στοιχείο GDAs και ε, άλλα στοιχεία που ισχύουν στις σκανδιναβικέ χώρες ε, θα έλεγα είναι άλλη υπόθεση. Επιπρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιούνται εθελοντικά. Δεν τα απαγορεύουμε. Μόνο που αυτά τα συστήματα δεν θέλουν να είναι υποχρεωτική χρήση πανευρωπαϊκά. Διότι δεν γνωρίζουμε καθόλου αν κατανοούν και θα κατανοούν οι καταναλωτές αυτά τα στοιχεία. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη που δεν υπάρχουν σκοτεινοί σηματοδότες. Τι θα κατανα... καταλαβαίνουν αυτοί εκεί για τα χρώματα αυτά. Και μετά όσον αφορά την επισήμανση αυτή δεν είναι ε, η πιο εύλογη. Δεν έχουμε μη γη τρόφιμα στην ε, αγορά που να κυκλοφορούν. Λοιπόν, εδώ έχουμε και ως στόχο για κάποια προϊόντα την 40χρονη γυναίκα. Αν προσπαθούν καν κάποιοι με τις συνιστόμενες ε, recommended daily allowances, ε, συνιστόμενη ημερήσια ε, ποσότητα να αναφέρεται αυτή έχοντα σημείο αναφορά σε έναν ενήλικα να χρησιμοποιείται για παιδιά δεν είναι το πιο θετικό. Εξαρτάται και από το φύλλο και από την ηλικία η συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέτοιες αναφορές. Επιπρόσθετα, όπως είπα, είναι δυνατόν να αναφέρονται. Και δεν είναι ε, ε, θέμα του ε, κράτους μέλους ξεχωριστά ένα κράτος μέλος να έχει στη διακριτική του ευχέρεια δυνατότητα υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος. Όχι. Ο τομέας σε ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί εθελοντικά κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Και το κάνουν ήδη τώρα κάποιοι. Αυτό το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Και όταν αναφέρονται κάποια στοιχεία είναι πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Αν θέλουν ε, οι καταναλωτές ε, και αν θέλει ο καταναλωτής υποχρεωτικά να έχει μια χρωματική ε, ταξινόμηση των προϊόντων, τότε θα προσαρμοστεί η αγορά στη συνέχεια. Αν θέλει ο καταναλωτής να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μόνο που δεν θέλουμε να γίνεται ούτε υποχρεωτικά αυτό, ούτε για το GDA, ούτε για τα χρώματα των φωτεινών σηματοδοτών στα προϊόντα. Είναι μόνο για προϊόντα convenience ε, και εφαρμόζεται εκεί. Δεν υπάρχει καμιά επιστημονική τεκμηρίωση που να δικαιολογεί αυτό. Το ε, φάσμα ως διαχωριστική γραμμή, δηλαδή μεταξύ ενός χρώματος και άλλου χρώματος, το εύρος είναι τεράστιο καθώς επίσης ε, και όσον αφορά συγκεκριμένες ποσότητες από, ένα, από μια ουσία. Έχει μεγάλη διαφορά η συμπίκνωση, το μέγεθος της ε, ποσότητας. Και γι' αυτό είπα, τα τρία χρώματα δεν μπορούν ποτέ να καλύπτουν την πολυμορφία όλων των χρωμάτων της ε, ήριδας και δεν είναι δυνατόν να επαρκεστούμε σε τρία χρώματα. Εκείνο το οποίο είναι αποφασιστικό όσον αφορά το, ε, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των καταναλωτών Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά πανευρωπαϊκά ε, να χρησιμοποιείται αυτό. Εθελοντικά μπορεί να γίνεται αυτό. Ολοκληρώνω. Α συνειδητοποιήσουμε ότι φυσικά αυτό ο κανονισμό που θέλουμε να γίνει είναι υπέρ των καταναλωτών. Θέλουμε να βοηθήσουμε του καταναλωτέ να παίρνουν μια καλή απόφαση στην αγορά τροφίμων. Δεν είναι όμω θέμα μόνο καταναλωτών. Είναι και για την άλλη πλευρά. Για του παραγωγού τροφίμων, τι εταιρείε που παραγούν τρόφιμα. Θέλουμε να του δώσουμε μια απλούστευση νομικού πλαισίου, νομική ασφάλεια και βεβαιότητα και εναρμονισμό στην ενιαία εσωτερική αγορά. Να είναι υποφελή η πρωτοβουλία μα και για τι δύο πλευρέ, αμφίπλευρα. Θέλουμε και για του δύο να κάνουμε κάτι. Και μόνο τον μέσο καταναλωτή μπορούμε να έχουμε ως στόχο. Μόνο τον κανονικό τον θα έλεγα καθημερινό καταναλωτή. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ασθενείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια επισήμαση που θα αφορά όλα τα τρόφιμα και όχι τα αλκοολούχα ποτά στην Ευρώπη. Αυτό είναι το εύρο και αυτό είναι ο τρόπο προσέγγιση. Όλα λοιπόν νομίζω ότι έχουν με αυτόν τον τρόπο αναφερθεί. Χαίρομαι για τι συζητήσει διμερό μαζί σας. Πρόεδρε, παρότι έχει προχωρήσει ο χρόνο, θα ήθελα κάποιο από το Συμβούλιο να μπορέσει να παρέμβει. Έχουμε και εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Θα ήταν ενδιαφέρον σύντομα να ακούσουμε τι απόψει του Συμβουλίου, κατά πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίες στο Συμβούλιο σχετικά. Ευχαριστώ. Äh, Μάλιστα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Α ζητήσουμε λοιπόν από το Συμβούλιο και να μα πει κατά πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίε από πλευρά του Συμβουλίου. Η κυρία Έτβινσον είναι. Το βλέπω σωστά. Εσεί παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να σας εκθέσω τις απόψεις του Συμβουλίου. Ακόμα δεν έχουμε κρυσταλώσει βέβαια κάποιες ε, θέσεις, αλλά μπορώ να σας ε, ε, πω τα πιο σπουδαία σημεία πρώτα-πρώτα όσον αφορά το πόσο κατανοητή θα πρέπει να είναι η νόμοθέσεις που θα θεσπίσουμε. Θέλουμε να υπάρξει τελικά μια ευρεία συνένεση για να μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε κάποια κριτήρια μετρήσιμα. Κάποιοι ήδη μίλησαν για κάποιες γενικές προϋποθέσεις ε, νομίζω ότι όλοι μας ε, έχουμε ε, δει κάποιο προϊόν, έχει πέσει στα χέρια μας μια συσκευασία ακατανόητη. Όμως αυτό ποτέ δεν είναι αγώγιμο, ποτέ κανείς δεν μπορεί να προσφύγει με δικαστήριο κατά του παραγωγού για αυτό το λόγο. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε και σαν κριτήριο το μέγεθος των στοιχείων είπαμε για τα δύο χιλιοστά ε, δηλαδή είπαμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει ως κριτήριο το μέγεθος του μικρού γράμματος χ, του στοιχείου χ. Επίσης θα πρέπει να δοθούν αυστηρές οδηγίες σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία, δηλαδή τι θα πει κόντρα στα αντίθεση χρωματική μεταξύ του background και των γραμμάτων. Τώρα όσον αφορά το διατροφικό προφίλ, αυτό ακόμα και αν φαίνεται ε, πάρα πολύ βαρύ, θα πρέπει να θεσπιστεί κατά τρόπο υποχρεωτικό. Να υπάρχει ένα πίνακα σε μία θέση με όλε τι πληροφορίε και όπω είπαν πολλοί πληροφορίε, ίσω θα πρέπει να έχουμε ανά 100 γραμμάρια, ανά 100 ε, μιλιλίτρε ε, την αναφορά του κάθε στοιχείου, του κάθε συστατικού. Από ό,τι καταλάβαμε περισσότεροι ε, θέλουν να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες όπου βέβαια τα διατροφικά στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στο μπροστινό μέρος ή μπροστά πλάι. Τώρα, τι θα αναφέρεται από αυτά τα συστατικά. Ε, τα λιπαρά ή ζάχαρη, αλάτι, ε, πολύ ακόρεστα. Αυτή το Συμβούλιο προέκυψε ότι αν τελικά διαγράψει ένα κομμάτι της πρωτοβουλίας, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε ε, θα καταλήξουμε σε εκτεταμένη δυσανάλογη απαγόρευση. Κανένας βέβαια δεν θέλει να δει για ε, όλα αυτά, όλες αυτές τις ιδέε τη βιομηχανία να υπάρξει μια γενική απαγόρευση. Άρα θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερα το πώ τελικά θα εφαρμόσουμε την νομοθεσία που θα θεσπίσουμε. Μάλιστα. Πολλή δουλειά απομένει ακόμα για το Συμβούλιο. Σα ευχαριστούμε κυρία. Η πρόταση εδώ και δύο χρόνια είναι σχεδόν επί τραπέζης. 31 Ιανουαρίου 2008. Νομίζω επαρκές χρονικό διάστημα ήταν να ασχοληθεί κανείς με αυτό το χατοφυλάκιο. Λοιπόν, προθεσμία, διορία για τι τροπολογίε 9 Δεκεμβρίου. 12 το μεσημέρι τελική διορία. Μέχρι το Μάιο θα μπορούσαμε αυτό το σχέδιο να μπορέσει να έχει περάσει από την Ολομέλεια και να έχει εγκριθεί. 9 λοιπόν Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρία Ζόμερ για αυτή την έκθεση. Λοιπόν, 18.00 προτείνεται. Εντάξει, ε, τότε λοιπόν 9 Δεκεμβρίου 18.006 το απόγευμα και όχι 12 το μεσημέρι. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Περνάμε στο σημείο 13 τώρα της ημερησίας διάταξης. Ένα εξίσου μεγάλο σοβαρό ζήτημα ως χαρτοφυλάκιο. Επικίνδυνες ουσίες στο, στα ηλεκτρονικά και ε, ήδη και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Α, μάλιστα λέει του, είπαν ότι είναι αντίθετη η σειρά. Μόλις μου είπαν ότι η έκθεση Sonic θα είναι η πρώτη που θα εξεταστεί. Ασφάλεια εφοδιασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο. Έχει τον λόγο κύριε Σόνικ, παρακαλώ. Και όλοι οι αρμόδιοι για τα τρόφιμα που το βρήκαν τόσο ενδιαφέρον και θέλουν να συζητήσουν κάτι, να συζητήσουν εκτός της αίθουσας παρακαλώ, εκτός αίθους οι συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η κυρία Εύανς ζήτησε να υπάρξει μια αλλαγή σήμερα σε διάταξη. Dear friends, all... αγαπητοί φίλοι, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να συζητήσουν, να αποχωρήσουν και να συζητήσουν εκτός εθούσης υπάρχει μεγάλος χώρος, ε, ελεύθερος χώρος μπροστά από την αίθουσά μας, έξω από την αίθουσά μας. Thanks The to the uh, Και το Συμβούλιο για το επόμενο θέμα. Ε, παρακολουθείτε. Ε, η Σουηδική εκεί ομάδα. Εντάξει. Please, we want to listen to Okay. Καλό Παρακαλώ και να ακούσουμε τον συνάδελφο. Κύριε, Κύριε Σόνικ έχει τον λόγο λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Εύανς διότι δέχθηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στην ημερήσια διάταξη ούτως ώστε τώρα να παρουσιάσω το θέμα μου. έχω ως βάση, ως αφετηρία την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής το σχέδιο του του κανονισμού, το ώστε να παρασχεθούν κάποιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση προμήθειας προσφοράς αερίου για να αντικατασταθεί η οδηγία 2004 κάθετος 66 που επίσης προέβλεπε τα της ασφαλείας ε, ε, παροχής του, του, του φυσικού αερίου. Όμως τώρα πλέον δεν επαρκεί ε, αυτή η οδηγία, αυτό το νομοθέτημα, διότι τώρα έχουμε ευξημένου κινδύνου όσον αφορά τη διέλευση του φυσικού αερίου από κάποιε τρίτε χώρε. Τώρα το 25% της κατανάλωσης, ε, δηλαδή το 60% των όσων έχουμε προέρχεται από κάποιες εισαγωγέ. και ε, επομένως σε σχέση με τα άλλα ορυκτά καύσιμα έχουμε να κάνουμε με μεγάλη συμβολή στον αφορά του θερμοκηπίου ούτω ώστε τώρα να έχουμε ένα πολύ μικρό αποτύπωμα. Έχουμε επομένω αυτή, αυτήν εδώ την πρόταση τη Κομισιόν που εντάσσεται στα πλαίσια των ε, προτάσεων για το 2020. και επομένως θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τη ζήτηση και ταυτόχρονα όμως να συνδυαστεί προ του με την ασφάλεια της ε, προσφοράς και στην Ευρώπη η ενέργεια να προέρχεται από βιώσιμες ε, πηγές και να μπορέσουμε να πάρουμε υπόψη τι υπάρχουσε ανάγκες. Και να κάτσουμε και να σκεφτούμε επίση ποιε είναι οι επιπτώσει πάνω ή στο περιβάλλον. Δεύτερον, θα πρέπει να μετακινηθούμε προς τα ορυκτά καύσιμα ε, λένε μερικοί, το οποίο όμως αυξάνει τις εκπομπές του διοξιδίου ε, ή να αντικαταστήσουν το φυσικό αέριο με άνθρακα ή ε, πετρέλαιο ή μαζούτ. Όμως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το να αποφεύγουμε κάποιες καταστάσεις κρίσης. Άρα θα πρέπει τα της ορθολογικής κατανάλωσης να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε την, ε, την τοπική διάσταση των ενεργειακών αναγκών και να χρησιμοποιούμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα παροχής φυσικού αερίου. Όμως ε, για να έχουμε σωστή υποδομή θα πρέπει να έχουμε πρώτα-πρώτα μία μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. να λάβουμε υπόψη τα του φυσικού περιβάλλοντος, τα, της προστασίας των πτηνών κλπ. Να λάβουμε υπόψη επίσης κάποια εθνική κληρονομιά και έτσι να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς ε, κάποια αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτός ο οργανισμός θα δώσει μια νέα όθηση στα 27 κρατημέλια αλλά και στις χώρες του ΕΟΧ. Άρα σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Πρώτη 12 του 2009. Και η συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ. Το δε άρθρο 194 της συνθήκης ορίζει ότι η ενεργειακή ελεγγύη είναι μια υποχρέωση. Επομένως τώρα έχουμε μια νέα, μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει αυτό το σχέδιο κειμένο. Να πρέπει να βλέπουμε μπροστά, όχι πίσω. Εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα και έτσι και σας προτείνω να κινηθούμε. Η δε συνθήκη της Λισαβόνας μας παρέχει μια βάση για να κινηθούμε αλληλέγγυα όσον αφορά και την ενεργειακή πολιτική. Υπάρχουν απειλές προς ε, την ενεργή αλλά θα πρέπει να δώσουμε τις αρμοδιότητες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο ώστε να προβεί διαπραγματεύσεις για την, ε, για την προσφορά της ενέργειας σχέση με τις χώρες και θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι κονσόρτσια ιδιωτικών εταιριών που δεν ε, δεν, δεν, δεν, δεν υπήκουν ε, αναγκαστικά στις αρχές του κράτους όπου εδρεύουν. Να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε δυναμικοί και να έχει περισσότερες αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φερρυπίν. Να μπορεί να επιβάλλει κάποια κατεπήγοντα μέτρα. Και παραλλήλως να υπάρχει ένα σχέδιο δράση για τέτοιες καταστάσεις, αλλά να μπορούμε να δράσουμε, να και προληπτικά. Είναι η περίπτωση σε κάποιο κράτο μέλο υπάρχει κατάσταση κατεπηγούσης ανάγκης. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιε καταστάσει που περιγράφονται και επομένω θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι διαφορετικέ καταστάσει, να έχουμε ιδιαίτερη ευελιξία και θα πρέπει κάθε φορά να, να, να, να, δούμε σε τι βαθμό κατεπήγοντο πόσο σοβαρή είναι μια κατεπήγουσα κατάσταση και πόσο θα διαρκεί. Όμω προσοχή, διότι πολλέ φορέ ε, έχουμε καταστάσει όπω τον Ιανουάριο τον περασμένο που είχαμε διακοπή τη προσφορά. Και ακόμα ένα κράτο μέλο αντιμετωπίζει προβλήματα από τότε. ούτε μπορούμε να πούμε ότι ακόμα έχουμε πλήρη απελευθέρωση του συστήματος ενέργειας, αλλά χρειάζεται να εξασφαλιστεί η προσφορά της ενέργειας. Θα πρέπει. όσο αφορά τι ε, υποδομές. Αν είναι δυνατόν να υπάρξει αντιστροφή τη ροή του φυσικού αερίου. Όμως, αυτό δεν δικαιολογείται οικονομικά. Πολλέ φορές δεν, δεν έχει νόημα το να αντιστραφεί η ροή. Τουλάχιστον για τι χώρε που παράγουν φυσικό αέριο. Άρα είναι θέμα ορθής απόφαση των ε, αρμοδιών αρχών σε κάθε χώρα μέλος ή από τα συντονισμένα όργανα ε, εδώ στο κέντρο στις Βρυξέλλες, παρά μόνο όταν υπάρχει τεκμήριος οικονομική. Τώρα, εγώ έρχομαι σε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρει λόγου. Πρώτα-πρώτα, διότι θέλω να υπάρχει καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τι ενεργέ μα. Δεύτερον, ε, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωτική ε, προσέγγιση με πρωτοπόρα ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προσφορά ενέργειας σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να συνδυαστεί η εξασφάλιση της ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος, ούτως ώστε η, παρεχόμενη στην Ευρώπη ενέργεια να είναι σύντονη με την αρχή της ε, βιωσιμότητας. Και εν τέλει παρακαλώ και εσείς να επιψηφίσετε αυτό το κείμενο. Σε ευχαριστούμε κύριε Σόνικ για αυτό το σχέδιό σας. Οι περιβαλλοντικές πτυχές αναφέρονται που για την δική μας Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Κρίς Ντέιβις πρώτος, παρακαλώ, Ντέιβις. Um, Στο Πρόεδρε, μου άρεσαν τα σχόλια του εισηγητή μία σκέψη. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ αυτή την έκθεση, αλλά το θέμα των εφοδιασμού της ενέργειας το παρακολουθώ και την ε, πρόθεση της ε, τεχνικής ε, συλλογής και αποθήκευσης του άνθρακα για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της χρήσης των ρηκτών καυσίμων. δεν υπάρχουν όμως κέντρα για να επενδύσουμε σε αυτή τη νέα τεχνική ή στα πυρηνικά ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, βλέπω σε μεγάλο βαθμό ότι ο κλάδος χρησιμοποιεί πολύ κόσμο για να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές. Αλλά στην πραγματικότητα ε, ο κλάδος επηρεάζεται βραχυπρόθεσμα. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα όλοι ζητάνε φυσικό αέριο. Όλοι αυτό ζητάνε, όλοι αυτό ψάχνουν. Παρά τις επιπτώσεις στον ανεφοδιασμό της ενέργειας. Φυσικά συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το φυσικό αέριο σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα, ε, τον άνθρακα και το πετρέλαιο, έχει χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αν όμως ε, θέλουμε να μειώσουμε μέσα σε 40 χρόνια κατά 80% τις εκπομπές μας ε, διοξιδίου του άνθρακα, σε κάποια φάση ε, κάπως αυτό, το διοξείδιο του άνθρακα που θα παράγεται από τι εγκαταστάσει ε, διοξείδιο του άνθρακα ε, κάπου θα πρέπει να αποθηκεύεται. Και οι μελλοντικέ εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν τέτοια συστήματα ε, και αποθήκευσης του διοξείδιου του άνθρακα. Τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν χώρο, αρκετό χώρο, ούτω ώστε ε, στο μέλλον κάποια στιγμή να ε, κατασκευαστούν και τέτοιες εγκαταστάσεις. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον άνθρακα ε, για να παράγουν ενέργεια θα πρέπει να βρουν και χώρους αποθήκευσης του του άνθρακα και με ε, τρόπους αποθήκευσης από τα εργοστάσια παρασκευής ενέργειας προς τα εργοστάσια αποθήκευσης του του άνθρακα. σε εγκαταστάσεις μάλλον αποθήκευση διοξύτου άνθρακα. Αυτά και ευχαριστώ τον εισηγητή για τα σχόλιά του. Ευχαριστώ. Κάποιες λίγες παρατηρήσεις και εγώ όπως ε, στα όσα είπε ο συνάδελφος. Ο προηγούμενος χειμώνας δείχνει ότι είναι κατεπήγον αυτό το θέμα και πρέπει να το λύσουμε. Είναι σαφές αυτό και ας είμαστε ειλικρινεί. Η μόνη πραγματική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η χρήση λιγότερου φυσικού αερίου. Αυτό θα πρέπει να είναι η επικέντρωσή μας, η εστίασή μας. Γενικά συμφωνώ με τον κύριο Σόνικ και τις απόψεις του. Τον ευχαριστώ για τη διατύπωσή τους. Υπογραμμίζω τη σημασία της έμφασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αηφορίας, απο, αποδοτικότητα στην εκμετάλλευση της ενέργειας όπως κάνει η Είμαι και στεναρά υπέρ τη ε, ρήτρα αλληλεγγύη ε, σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα που άρχισε να ισχύει σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε δυνατότητε αποθήκευση θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι περνάει από το χέρι τη όσο αφορά τι αρμοδιότητέ τη, ώστε η προσπελασιμότητα, η προσβασιμότητα σε τέτοιου είδου ε, εγκαταστάσει αποθήκευση ε, να είναι εφικτή. Τώρα, δεν συμφωνώ σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Μια στιγμή να το βρω. Για τον στόχο 2014 για τις αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν σε σχέση με μια διακοπή όσον αφορά την υποδομή, να, αν να υπάρχει η ε, δυνατότητα να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Είναι έντονη η ανάγκη μας ε, να εφοδιαζόμαστε με φυσικό αέριο. Πρέπει τα μέτρα αυτά να ληφθούν άμεσα. Το να περιμένουμε μέχρι το 2016 θα είναι υπερβολικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γιάννος Άντερ. Έχω δύο ερωτήματα. Ίσως δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος να τα θέσω και ίσως δεν θα πρέπει να τα απευθύνω στον κύριο Σόνικ. Αλλά από το υλικό που έχουμε ε, δεν παίρνω απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και θα τα θέσω. Ο κύριος Σόνικ ανέφερε ότι υποστηρίζει έντονα το, το σύστημα εφοδιασμού θα πρέπει να είναι κατάλογος, ε, κατάλληλο, ούτω ώστε να υπάρχει και αντιστροφή της ροής του αερίου σε λίγα χρόνια. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό δικαιολογείται. Όσοι όμως το καταλαβαίνουν, λένε ότι αυτό θα κοστίσει απίστευτα λεφτά για να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα μπορεί να αντιστρέψει τη ροή του φυσικού αερίου. Έχει υπολογίσει κανείς το κόστος αυτής της αντιστροφής. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο αφορά και πάλι χρήματα. Μιλάμε για τα, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που θα πρέπει να φτιάξουμε. Ε, θα πρέπει να είναι παρκής για 60 μέρες ε, με το χειρότερο σενάριο του πολύ δρυμή καιρού, ας πούμε. Έχει κάνει κανένα υπολογισμό πόσο θα μας κοστίσει να έχουμε τέτοιες τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Στο υλικό που μας δώσατε δεν έχω βρει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να μου δώσετε απάντηση αν μπορείτε παρακαλώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Γιούστα Παλέτσκης παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω εγώ ότι όπως πιστεύω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε, συνέταξε ένα καλά διατυπωμένο έγγραφο. Και όσον αφορά τη γνωμοδότηση από πλευράς του κυρίου Μπόγουσλαου Σόνικ, είναι πάρα πολύ καλή και θα βοηθήσει αυτή η γνωμοδότηση του κυρίου Σόνικ να βελτιωθεί αυτό το έγγραφο ως πρόταση. Να αναφέρω κάποια σημεία επιπρόσθετα εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να διευρύνουμε την, το πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας. Ιδιαίτερα για μικρές χώρες μόνο περιφερειακά τοπικά προγράμματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών μπορούν να είναι λειτουργικά για να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά έκτακτης ανάγκης, π.χ. βαλτικές χώρες. Εδώ θα μπορούσε να αναλάβει ιδιαίτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συντονισμό και την διευκόνιση αυτής της περιφερειακής διασυνοριακής συνεργασίας. Ιδιαίτερα και όσον αφορά και άλλες χώρες, όχι μόνο στη Βαλτική και για τις νέες χώρες επίσης πιστεύω επίσης για την ευθύνη να αυξηθεί η δυνατότητα διασύνδεσης σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επικοδομητικός και ο ρόλος των διαθετικών των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Επίσης σε όλα τα ε, προγράμματα για τις υποδομές όταν έχουμε μια κατάσταση έκταξη ανάγκης, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά καύσιμα, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις πάντα. Τώρα για την περίπτωση ορισμού των προστατευόμενων πελατών ή καταναλωτών, συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Σουονιεκ ε, εισηγητού να μείνει ανοιχτός αυτός ο κατάλογος. Όμως όσον αφορά τα νοικοκυριά υποθέτω θα πρέπει να αναφέρουμε όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχολεία και νοσοκομεία, κλινικές, αλλά επίσης ε, και άλλους τομείς ε, ευάλωτους όσον αφορά την παροχή δημόσιων κρατικών υπηρεσιών, όσον αφορά νηπιαγωγία, για παράδειγμα ορφανοτροφία και γυροκομεία. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόνικ τώρα θα ήθελε να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, λέει η κυρία Μουρκουνάιτε, καλωσορίζω την γνωμοδότηση και ευχαριστώ και τον κύριο Σόνικ για τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε για να ετοιμάσει το έγγραφο. Αυτά που λέει το κείμενο για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και μια μελέτη αντικτύπου για το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικά, ειδικά ε, για μεγάλα προγράμματα επενδυτικά. Ε, ξέρω περιπτώσεις ε, μεγάλων τέτοιων προγραμμάτων που δεν έγινε τέτοια μελέτη αντικτύπου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη ροή του φυσικού αερίου την απρόσκοπτη ροή του φυσικού αερίου και να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλοι μας εξαρτώμαστε από ένα και μόνο προμηθευτή, τη Ρωσία. Και με βάση τα νέα που έχουμε από την Χάγη χθες, ε, δείχνουν ότι η Ρωσία δεν ακολουθεί, δεν σέβεται τον ενεργειακό χάρτη. Και ότι θα χρειαστεί να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο για την παραβίαση της χάρτας. Ε, Ευχαριστώ κύριο Σόνικ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις του κυρίου Άντερ για το κόστος των υποδομών. Έχει γίνει και το αν έχει γίνει αξιολόγηση του κόστους. Κανονικά η Κομισιόν θα πρέπει να μας απαντήσει. Ε, από ό,τι ξέρω η Κομισιόν έχει κάνει τέτοια αξιολόγηση. Ε, έχει εκτιμήσει το κόστος ε, της ε, αντιστροφής των ε, ροών του φυσικού αερίου και δεν είναι πολύ ψηλό από ό,τι ακούω. Ε, και μάλιστα προβλέπονται και κάποια κοινοτικά κονδύλια για να υποστηριχθούν αυτού του είδους υποδομές. Τώρα, γιατί περάσαμε στην ημερομηνία του 2016, γιατί θα πρέπει οι σχετικές υποδομές τότε να είναι έτοιμες σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν που είχε προβλέψει το 2014. Γιατί θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Ο συνάδελφος από τη Λιθουανία είπε ότι χρειαζόμαστε αξιολογήσεις ε, αντικτύπου στο περιβάλλον. Συχνά αυτές οι αξιολογήσεις, αυτές οι μελέτες είναι χρονοβόρε. Και πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να ετοιμαστούμε. Ακριβώς γι' αυτό πρότεινα αυτή την ημερομηνία. Για τον Nord Stream. Το Nord Stream έχει ετοιμάσει μια μελέτη αντικτύπου δεν θέλω να μιλήσω για την ποιότητα της μελέτης αυτής, αλλά χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να ετοιμάσω αυτή τη μελέτη. και προέκυψε τέλος πάνω, μία εκτίμηση από αυτή τη μελέτη. Προς τον κύριο Ντέιβις. Ναι, θέλω ε, καθαρές τεχνολογίες άνθρακα. Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τον άνθρακα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Η Πολωνία παράγει τέτοια ενέργεια. Κατά 90% της ενέργειά μας βασίζεται στον άνθρακα, παράγεται από άνθρακα. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτά τα συστήματα ε, με το σύστημα δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα και να βρούμε κάποιες λύσεις για το πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το διοξίδιο του άνθρακα για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Νομίζω ότι είναι θέμα των κρατών μελών. Αυτά θα αξιολογήσουν αν χρειάζεται να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια στα κράτη-μέλη. Ε, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν. Η Κομισιόν δεν μπορεί να επιβάλλει ε, τέτοιο, κάτι τέτοιο στο κρατός μέλος και να επιβάλλει οικονομικό άχθος. Ε, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για να ετοιμάσει ένα σχέδιο κατεπήγοντος σε περίπτωση που υπάρχει έλλειμμα ενέργειας. Ο κ. Παλεύσκη έχει δίκιο. Θα χρειαστούμε τέτοια σχέδια κατεπήγοντα σε περίπτωση που υπάρχουν απειλές για τη ροή της ενέργειας στην περίπτωση που υπάρχουν διαταραχές, φυσικά χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις. Εγώ έχω κάνει κάποιες ε, υποδείξεις, κάποιες προτάσεις για το σημείο ακριβώ αυτό. Και φυσικά θα πρέπει να σκεφτούμε και τις ανάγκες των ε, πολιτών μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά. Οι, τους που επιτελούν δημόσιο έργο, όπως παραδείγματος χάρη τα ορφανοτροφία, η... τα νηπιαγωγεία, η... τα γυροκομεία, τα οποία θα μπορούσαν να πληγούν πρώτα και καλύτερα σε περίπτωση κρίσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σόνικ για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Σημαντικό ζήτημα η έκθεση αυτή. Χωρίς ανεφοδιασμό ενεργειακό η ζωή μας δεν θα ήταν δυνατόν να είναι ευχάριστη. Αναφέρθηκαν οι περιβαλλοντικές πτυχές και φυσικά και τα κόστη σε σχέση με αυτές τις πτυχές που πρέπει να τα δούμε. Προτείνουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών πάλι 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Εντάξει, για την έκθεση Σόνικα αυτή η προθεσμία. Και περνάμε στη συνέχεια στο τελευταίο σημείο για απόψε. Έκθεση Florence του κυρίου Φλωρεντίου για σωστό λάθος. Τι λέτε μια ματιά στην ημερήσια διάταξη διευκολύνει την διαπίστωση της σειράς. Είμαστε στην έκθεση Jill Evans μάλιστα αυτή για τους περιορισμούς στην χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών ε, στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ε, αναδιατύπωση της πρότασης. Ο κύριος Evans. Thank you very much, uh, Κυρία Εύαν, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το προηγούμενο μήνα και είχαμε και μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι όλοι είχαν την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στην έκθεση. Είναι σημαντικό, θα έλεγα, πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε το εύρος του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε εδώ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε ε, έχουμε 9 εκατομμύρια τόνους ε, ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρικών συσκευών που οι περισσότερες από αυτές ε, είναι ε, τηλε, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εξοπλισμός νοικοκυριών. Αυξάνεται 200 και με αυτά τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών βλέπουμε επιτάχυνση των, του όγκου και εκτιμάται ότι το 2020 θα έχει αυξηθεί σε πάνω από 12 εκατομμύρια τόνους. Το να πρασινίσει αυτό λοιπόν, να γίνει πιο φιλοπεριβαλλοντικό αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό διότι μπορεί να έχει βλαπτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία αν δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα απόβλητα σωστό, σωστά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναψώμενες χώρες. Και σύμφωνα και με την συνθήκη, η περιβαλλοντικές ζημιές θα πρέπει στην πηγή τους ε, να επαναρθώνται, να θεραπεύονται. Επίσης έχουμε και προτεραιότητα στον τομέα της πρόληψης, δηλαδή μείωση των ε, βλαπτικών ουσιών όσον αφορά τα προϊόντα αυτά και την χρήση τους. Η οδηγία που υιοθετήθηκε το 2003 βασιζόμενη σε μια πρόταση του 2000 ήθελε με μια κλιμακούμενη διαδικασία να αντιμετωπίσει βαρέα μέταλλα και άλλες λαπτικές ουσίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε σε μείωση κατά πάνω από 100.000 τόνους αυτών των ε, ε, υλικών. Και ενώ είναι σημαντικό όχι μόνο θέτοντας ευρωπαϊκές προδιαγραφές αλλά και παγκόσμιες προδιαγραφές ε, δεν έχει παρακολύσει την περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων και είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Επανασχεδιάστηκαν προϊόντα ώστε να συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες και μάλιστα έχουν ξεπεράσει και αυτό το πλαίσιο και όσον αφορά και την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης αντικατάστασης. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και φαίνεται ότι από τις συζητήσεις που είχαμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων να διευρυνθεί το εύρος της οδηγίας ώστε όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές να καλύπτονται και όχι μόνο κάποιες κατηγορίες αυτών. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος νομίζω που θα μπορούμε να έχουμε νομική βεβαιότητα, νομική ασφάλεια αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι άπαντα τα προϊόντα πρέπει να καλύπτονται από αυτή την οδηγία, διότι προτείνει κάποιες εξαιρεσει από αυτό το πεδίο εφαρμογής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορώ με κάποιες ε, προϋποθέσεις να δεχθώ αυτές τις εξαιρέσεις. Τώρα, σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο θέματα κλειδιά. Το ένα είναι έναντι του ε, REACH όσον αφορά το ε, ROSH έναντι του REACH των χημικών δηλαδή ουσιών όσον αφορά το ΡΟΣ. Αυτό τι σημαίνει σε σχέση με τις ε, εξαιρέσεις ε, μέσα σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. Θα πάρει πάνω από μια δεκαετία για την πλήρη εφαρμογή και δεν θα αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα των κυριότερων ουσιών που δημιουργούν τα προβλήματα σε σχέση με την οδηγία ΡΟΣ το PVC και οι επιβραδυντές σε σχέση με την πυρκαγιά βρωμιούχα κτλ και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε αυτές τις ε, σύνθετες ουσίες ε, και την ε, αδειοδότηση και αξιολόγησή τους. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο του ΡΟΣ και δεν είχε σχεδιαστεί έτσι και ελπίζω ότι θα συμμεριστεί τις απόψεις μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θεωρούν το ΡΟΣ συμπληρωματικό στοιχείο του «ΡΙΤΣ» και με αυτόν τον τρόπο και από πλευρά τη ε, υπηρεσία ε, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών Ουσιών προσεγγίζεται. Θα ήθελα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δούμε την οδηγία για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος και να μην αντικαταστήσουμε αυτό με κάτι άλλο που δεν θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα καθόλου. Το δεύτερο σημείο κλειδί είναι οι νέοι περιορισμοί και θα ήθελα αυτό κάπως πιο λεπτομεριακά να το δούμε νομίζω είναι το πιο επίμαχο θέμα, το πιο αμφίσιμο ζήτημα το οποίο συζητούμε. Το 2003 το άρθρο 6 Ρος υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά και κατηγορηματικά να εξετάσει την, το εφικτό της αντικατάστασης των επικίνδυνων ουσιών και να υποβάλει νομικές, νομοθετικές προτάσεις να διευρυνθεί το πεδίο του άρθρου 4, αν αυτό είναι ενδεδειγμένο. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαγραφεί αυτό το άρθρο και ανταυτού να εξεταστούν νέοι περιορισμοί υπό τη διαδικασία επιτροπολογίας υπό μια διαδικασία που θα σχεδιαστεί από πλευράς επιτροπολογίας. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη διεργασία και μάλιστα να χάναμε τη συναπόφαση εμείς ως Ευρωβουλή διότι το ΡΟΣ είναι συγκεκριμένα για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών και πιστεύω ότι θα έπρεπε να διατηρήσουμε τις δικές μας εξουσίες και αρμοδιότητες ως Ευρωβουλή για αυτό το θέμα. Πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν τη συζήτηση στο τι θα έπρεπε τώρα να κάνουμε άμεσα και όχι για το τι θα μπορούσε να γινόταν στο μέλλον ή κάποτε υστερότερα. Και αυτό νομίζω είναι η ευκαιρία που μας προσφέρεται στην οδηγία αυτή με τη νέα ρήτρα που στόχο είχε να διευκολύνει την δράση και όχι να αναβάλει ή να παρακολύσει ανάληψη δράσης. Προτείνω λοιπόν την επέκταση της απαγόρευσης σε τέτοιου είδους υλικά κατά, για 3,5 χρόνια μετά την έναρξη σε ισχύ της αναδιατυπωμένης αυτής πρότασης. Και για την ε, αιτιολογική σκέψη και το επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο χρησιμοποίησα για να επεξηγήσω τα κυριότερα επιχειρήματα όσον αφορά τις, ε, ε, τους περιορισμούς. Εδώ έχουμε τρία παραστοιχεία. Πρώτον, τεκμήρια για τις αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τα αλογονούχα και τους επιβραδυντές φλόγας. Και εδώ σε σχέση με τα βρωμιούχα υπάρχουν όμως πολλά άλλα τα οποία θέτουν τα ίδια προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποτιμήσει και να αξιολογήσει αυτές τις ουσίες. Αυτή η μελέτη λοιπόν ε, έδινε σύσταση ώστε η οργανοβρομεΐνη να μπορέσει να αντικατασταθεί όσον αφορά τις βλαπτικές της επιπτώσεις και για τους επιβραδυντές φλόγας και για να μπορέσει και, ακόμα και σε μονάδες αποτέφρωσης ε, να αντικατασταθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά την προηγμένη αντιμετώπιση αποβλήτων. Αυτές όμως οι εγκαταστάσεις ε, και διευκολύνσεις δεν υπάρχουν ούτε καν στα κράτη-μέλη, για να μην κάνουμε καν λόγο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι το SOPS. Στην πηγή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα Υπάρχει και ένα θέο, δεύτερο πρόβλημα με τους επιβραδυντές ε, φλόγας ε, όσον αφορά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας ε, και όσον αφορά και τις επιπτώσεις τους με την κλιμακούμενη αντικατάσταση μπορούμε και να ευθυγραμμιστούμε όσον αφορά και την χρήση των πλαστικών και είμαι βεβαία ότι θα έχουν έρθει σε επαφή οι συνάδελφοι θα τους έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους οι εταιρείε παραγωγή ή άλλες ενώσεις παραγωγών σε σχέση με τους κυριότερους λογονούχους και βρο... φλόγα φλόγας που χρησιμοποιούν βρωμιούχα προϊόντα και θα τους είπαν ότι δεν είναι τόσο ε, επικίνδυνα. Όμως ε, αυτό μας ε, κάνει να πούμε ότι περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής ε, και το πεδίο κινδύνων υπάρχουν και για παράδειγμα κοίταξαν μόνο τις ε, άμεσες ε, επιπτώσεις όσον αφορά την φάση αντιμετώπισης των αποβλήτων και όχι και το θέμα της ανακύκλωσης των πλαστικών ουσιών και των συνθετικών. Και φαίνεται ότι τα TBBPA που εμπεριέχονται σε αποτεφρωτές υψηλής θερμοκρασίας είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα συναφή θέματα που αφορούν και την δημιουργία πρόκληση διοξινών και αυτά τα οποία παρατηρούνται πολλές φορές και σε χωματερές. Αυτά τα θέματα αναφέρθηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν διότι δεν μπόρεσαν να ποσοστοποιηθούν οι όγκοι υλικών που χρησιμοποιούνται εκεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ακόμα και με τους περιορισμούς ε, της αποτίμησης κινδύνων, η πραγματική κίνδυνη της δημιουργίας διοξινών όπως καταδείχθηκε στη μελέτη και τα προβλήματα που προκαλούνται σε σχέση με την ανακύκλωση το θέμα της αντικατάστασης ε, των βρωμιούχων ε, επιβραδυντών ε, φλόγας είναι ένα ζήτημα και σε σχέση με το PVC και για τη μελέτη που ζητήθηκε να συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δόθηκε σύσταση ότι τα PVC πρέπει να αντικατασταθούν. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που αφορά απόβλητα PVC γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επεξηγηματική πρόταση γι' αυτό από το 2000 αναφέρει ότι υπάρχει επαρκής, ε, υπάρχουν επαρκή τεκμήρια ότι το PVC δεν είναι υλικό κατάλληλο για αποτέφρωση, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο και τον επικίνδυνο χαρακτήρα των υπολοιμάτων, ιδιαίτερα και όσον αφορά και τις ε, πλαστικές ουσίες και τις επιπτώσεις τους όσον αφορά χωματερέ ε, και με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ λίγα απόβλητα PVC αυτή τη στιγμή ανακυκλώνονται. Δυστυχώς αυτά τα τεκμήρια υποβλήθηκαν πολύ αργά για να συμπεριληφθούν στο ΡΟΣ τότε και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ε, θεωρήσουμε ότι ε, επαρκούσαν. Δεύτερο σημείο, η δράση όσον αφορά τους ε, παραγωγούς. Η ε, ηγετικοί κύκλοι όσον αφορά τους παραγωγούς βρίσκονται πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς. Έχουν αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή ε, χρήσεως αλογονούχων και την αντιμετώπιση των PVC και υπάρχει μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπέρ του περιβάλλοντος όσον αφορά την Παγκόσμια Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Δεν κάνουν λόγο για το αν θα έπρεπε να γίνει αυτή η ε, διαδικασία, αλλά για το πότε και με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει. Και αν η ίδια η βιομηχανία ηλεκτρονικών με τόσο σύνθετα περίπλοκα προϊόντα που παράγει μπορεί να οδηγηθεί στην χρήση χαμηλών αλογονούχων τα επόμενα χρόνια, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα για ε, τον άλλο τομέα να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς, ε, ώστε να μπορέσουμε, για παράδειγμα, να αποφύγουμε την χρήση PVC στα, ε, στα ψυγεία. Το άλλο στοιχείο είναι οι πρόσθετες ουσίες. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν να αποφασίσουμε για περαιτέρω περιορισμούς ε, για τους αλογονούχους ε, επιβραδυντές ε, φλόγας. Και τέτοιου είδους πληροφορίες όμως είναι διαθέσιμες. Δεν είναι το ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μας. Um, Ένας άλλος, ένα άλλο στοιχείο που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη είναι το ότι δεν υπάρχει παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιβραδυντών ε, φλόγας αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, τέτοια επικίνδυνα ε, παράγωγα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτίθενται σε αυτά χιλιάδες εργαζόμενοι. Επίσης ε, βλέπουμε ότι και για τις εναλλακτικέ ουσίες έχουμε μεγαλύτερους παραγωγούς. Δεν κάνουμε λόγο λοιπόν ε, για την πάυση λειτουργίας μιας ε, βιομηχανίας, αλλά για μια μετάθεση δραστηριοτήτων για την παραγωγή πιο ασφαλών ουσιών. Εδώ δεν τίθεται το θέμα της αμφισβήτησης πιο ασφαλών ουσιών, τίθεται όμως το θέμα κόστους. Αν ξαναδούμε όμως το θέμα κόστους και σε σχέση με την εναλλακτική δυνατότητα για το PVC και το ε, κόστος αυτό δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα ήταν μικρό. Ολοκληρώνω πρόεδρε. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται στην πηγή τα περιβαλλοντικά προβλήματα, στην πηγή όπου προκαλούνται. Και αυτό ήταν και αρχική πρόταση Ρος είναι η παραγωγή ε, προϊόντων χωρίς την χρήση καδμίου και άλλων βαρέων μετάλλων. Τώρα πρέπει να έχουμε τις ευκαιρίες συνεργαζόμενοι με τη βιομηχανία για την παραγωγή της νέας γενεάς ε, εξοπλισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ε, συσκευών χωρίς PVC και χωρίς επιβραδυντές φλόγας. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Evans για αυτή την μεσθένος ε, συνταχθήσα και παρουσιαστήσα έκθεση. Περνάμε τώρα στη φάση της συζήτησης. Οι σκιώδεις εισηγητές θα έχουν τον λόγο. Ο κύριος Μπόκουσλαβ Σόνιεκ λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ήβανς για την έκθεσή της. Ευχαριστώ και για όλες τις συνεδριάσεις που με βοήθησαν να διαμορφώσω γνώμη. Μία επέκταση του πεδίου της οδηγίας για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλές επιπτώσεις στο περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και θετικές επιπτώσεις στην οικονομία. Θα πρέπει να επεκτείνουμε το κείμενο αυτό σε όλους τους τομείς α, ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρικών συσκευών. Έχω παρόλα αυτά κάποιες α, ανησυχίες για τις νέες ουσίες που θα πρέπει να περιοριστούν. Εσείς αναφερθήκατε στο PVC στα βρωμιούχα και στους βρωμιούχους και χλωριούχους επιβραδυντές φλόγας. Θα πρέπει ε, να έχουμε ουσίες ούτως ώστε οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρικούς, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές ε, συσκευές με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το θέμα είναι ότι τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ε, συσκευών μπορούν οι κατάλληλοι φορεί να τα επεξεργαστούν. Έχουμε στοιχεία ότι αυτές οι ουσίες είναι τόσο επικίνδυνα για να αντικατασταθούν. Επίσης, δίνουμε 3,5 χρόνια για την αντικατάστασή τους. Νομίζω ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι υπερβολικά σύντομο. Θα πρέπει να συζητήσουμε πιο πολύ με τα κράτη-μέλη τη χρονική περίοδο για την αντικατάστασή τους. Το θέμα της ε, απαγόρευσης της ε, χρήσης των ουσιών, της παράλληλης απαγόρευσης, ε, αν έχω μια γενική απαγόρευση, θα οδηγηθούμε στη χρήση υποκαταστάτων που δεν έχουν αποδείξει ότι είναι λιγότερο επικίνδυνες και δεν νομίζω ότι θα προστατεύσουμε έτσι τους καταναλωτές και θα περιορίσουμε και την μόλυνση. Πώς, πώς θα γίνει κάτι τέτοιο αφού δεν έχουμε δοκιμάσει τις νέες ουσίες. Τώρα, για τις εξαιρέσεις από την ε, οδηγία. Θα πρέπει να είναι μια μεταβατική λύση ε, καθοδόν προς πιο φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τις ε, μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις. Ε, το REACH μας βοηθάει για να επιμεριστούν τα κόστη, κάτι που ευνοεί τις μικρές επιχειρήσεις. Τέτοιες δράσεις βοηθούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε τα μονοπόλια στην αγορά. Στο σημείο 13 του προημίου τροπολογία 10, κάτι τέτοιο γίνεται δυνατόν. Ε, δηλαδή, μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ληφθούν υπόψη εάν δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που υποδεικνύουν προς τη χρήση ενός υποκατάστατου. Για τις τροπολογίες 38 και 39. Αν οι τροπολογίε αυτέ δεν μα επιτρέψουν να βάλουμε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, πώ θα προχωρήσουμε. Στην τροπολογία 16 μιλάμε για τον ε, ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα πρέπει να είναι ασφαλή και αξιόπιστο. Επίση, ο εξοπλισμό στου πυράβλου, στην αεροπορία, στου δορυφόρου κτλ. Ε, Επίσης, ο χρόνο που χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά υλικά στι μεταφορέ είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στα νοικοκυριά. Ε, εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας των επιβατών. Ε, είσαστε σίγουροι ότι η τεχνολογία χωρίς μόλιδο είναι αρκετά ασφαλής. Ε, είσαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και αξιόπιστες και ασφαλείς μεταφορές έτσι και μεταφορές που κινούνται με ταχύ ρυθμό. Μεταφορικά μέσα που κινούνται με ταχύ ρυθμό. Τροπολογία 41. Ένας επιχειρηματίας λέγεται εδώ, θα πρέπει να φέρει το βάρος της απόδειξης. Ίσως θα πρέπει να έχουμε το σύστημα που ανέφερα πριν, δηλαδή του επιμερισμού του κόστους, όπως γίνεται στα πλαίσια του REACH. Και άλλα δύο σχόλια έχουμε να κάνω. Βεβαίω εν μέρει τα έχετε απαντήσει. Ε, πρότεινα στον εισηγητή να προσθέσει και μια γενική απαγόρευση για την ομάδα των βρωμιούχων ε, νόσεων, τροπολογία 70. Το θέμα είναι, έχουμε επιστημονικά στοιχεία υπέρ της απαγόρευσης. Εσείς αναφέρατε την μελέτη της Κομισιόν. Καλό θα ήταν να ακούσουμε διαστόματος επιτροπής την άποψή της για το θέμα αυτό. Mm, και στο τελευταίο μου ερώτημα, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι χημικές ουσίες. Ε, στους δρομιούχους επιβραδυντές φλόγας. Τι στοιχεία έχει ο εισηγητής για τις ε, αξιόπιστες εναλλακτικέ λύσεις, για, τις, ε, για τα υποκατάστατα αυτά. Αυτές οι, οι διαφορετικές ενώσεις είναι ασφαλείς και είναι εξίσου αποτελεσματικά τα μηχανήματα που τις χρησιμοποιούν. Σα ευχαριστούμε κύριε Σόνικ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει στο τέλος σε ερωτήματα σαν και αυτά. Τώρα η Κάτερίν θα έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ.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 θα πρέπει να δούμε το ότι όντω διαμορφώνεται μια συνένεση σε σχέση με το να περάσουν και οι δύο οδηγίε και ελπίζω ότι τέτοια συνένεση θα υπάρχει και στο Συμβούλιο. Διεύρυνση του πεδίου και έτσι να καλύψουμε ε, και τις ε, ηλεκτρονικές συσκευέ. Αυτό ε, το προτείνει και η συγκήτρια και θα την στηρίξουμε. Να δούμε τι θα γίνει με τις εξαιρέσεις και να δούμε τι θα γίνει με κάποιες κατηγορίες προϊόντων λοιπόν που ολόκληρες ε, εξαιρούνται αυτές εξ αρχής. Να δούμε θα γίνει και με αυτές τις, ε, τις υποχρεώσεις για απόσεις, για ανάκληση προϊόντος. και θα πρέπει να μας μιλήσει σχετικά η συγγήτρια. Και τι θα γίνεται επίσης με του, τα, τα ηλιακά πάνελ, αυτά τους θερμοσυσσωρευτές, τις συστοιχίες των θερμοσυσσωρευτών της ηλιακής ενέργειας. Και να δούμε τι θα προταθεί ε, σε σχέση με αυτό από την εισηγήτρια τώρα. Το πιο σημαντικό από αυτά τα οποία ε, συζητούνται, το πιο σημαντικό σημείο της έκθεσης είναι εκεί που αναφέρει συγκεκριμένα προϊόντα. Έχει εδώ ένα μεγάλο κατάλογο και απαρίθμηση στο τέταρτο παράρτημα. Ε, αναφέρει την πρόταση της Κομισιόν στο τέταρτο παράρτημα και επαναλαμβάνει κάποια πράγματα στο τέταρτο παράρτημα, όμως όσον αφορά τους επιβραδυντές φλόγας και εδώ έχει και διάφορες λέξεις που είναι πάρα πολύ να προφέρει κανείς και επίσης όσον αφορά το PVC. Πολύ φιλόδοξη πρόταση. Εμένα με βρίσκει σύμφωνη όμως και αξίζει της υποστήριξης όλων. Θα πρέπει ό,τι υποκατάστατα βρεθούν να είναι καλά μελετημένα, να είναι βιώσιμα και γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουμε για να δούμε ακριβώ πώς έχει η κατάσταση και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Και όπω προτείνει η συγκίτρια, να υπάρξει μια εκτίμηση του κινδύνου για τα διαφορετικά προϊόντα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε και εδώ θα πρέπει να μα πει η Επιτροπή τι πιστεύει. Δεν ξέρω αν θα προτείνει η Κομισιόν και άλλες ουσίες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συναπόφευση και όχι επιτροπολογία όσον αφορά την διαγραφή κάποιων προϊόντων ή ουσιών από το κείμενο. Σας ευχαριστούμε. Κρις Ντέιβις τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακόμα μια φορά ήταν κρυστάλλινη η έκθεση της ε, εισηγήτριας, αλλά θα πρέπει να τι θα γίνει με την, με την ε, του πεδιοφαρμογή. Είναι πολύ πράσινη αυτή η έκθεση, πολύ περιβαλλοντική. Συνήθω μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Δεν ξέρω όμω. Μπα και έτσι όμω δεν είναι τόσο ισορροπημένη. Γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορηματική όσον αφορά την απαγόρευση διαφόρων πραγμάτων. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε όχι κάποιο κάποια πρέπει να είναι επικίνδυνα από μόνο του, αλλά επειδή δημιουργούν κινδύνου. Άρα να είμαστε πιο προσεκτικοί στι απαγορεύσει. Γιατί το ότι θεωρητικά υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Ε, αυτό θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο. Θα πρέπει κανείς να αποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος και να απαιτείται αντικατάσταση προϊόντος με άλλο που θα αποδειχθεί ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι δεν θα υποστηρίξω την έκθεση, αλλά δεν με έχει πείσει 100% ότι αυτά τα οποία θα απαγορεύσει είναι τόσο επικίνδυνα, πραγματικά επικίνδυνα για περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Και ότι όλο αυτό προτείνει βιώσιμο και ασφαλή. Και αξιόπιστα και ότι θα λειτουργούν, γιατί μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λειτουργεί. Να δούμε τι θα μας πει και θα μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τώρα την έχουμε κάπως τριμώξει, ιδίω μια που η συγκέντρια εδώ αναφέρει κάποια μελέτη της Επιτροπής, που λέει, που, λέει πόσο πρέπει να απαγορευτούν οι επιβραδύντες φλόγας. Σαν ανακύκλωση υπάρχει πρόβλημα, με κάποιες από αυτές τις ε, ουσίες. Και άμα δεν γίνεται ανακύκλωση, τότε θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού τέλο πάντων. ως αφορά την ανάκτηση ενέργειας Διοξίνε δηλαδή. Οι διοξίνε που με αυτόν τον τρόπο αυθένονται στην ατμόσφαιρα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο αμφίβολα. Άρα, πού πάμε και για τα ηλεκτρονικά. Το θέμα είναι πώς θα θεσπιστούν, πώς θα χρησιμοποιηθούν κάποια, ε, κάποια υποκατάστατα, υποκατάστατες συσκευέ. Οι λομπίστες επιμένουν σε αυτό. Ίσως έχουν δίκιο. Ίσως αποδείξουν ότι θέλει κάποιες από αυτές τις αλλαγές ο κλάδος. Οπότε άμα θέλει, εντάξει, να προχωρήσουν προς τα εκεί. για το φωτοβολταϊκό τόξο. Ακούσαμε την άποψη των λόμπι. Τα πλεονεκτήματα για το περιβάλλον που λένε ότι θα έχουμε. Ότι θα έχουμε λένε 100% βελτίωση, καλύτερε επιδόσεις για ανακύκλωση κλπ. Και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για περιβάλλον ή για τον άνθρωπο. Να δούμε. Είναι έτσι. Αν είναι έτσι, τότε αυτή η νομοθεσία έρχεται μετά από έξι χρόνια αφού είχαμε την πρώτη σχετική νομοθεσία. Και άρα θα πρέπει σε έξι χρόνια να ξανακάνουμε κάτι μια που το ρίτς τότε θα τρέχει κανονικότατα. Άρα τι λέει η συγκεντρία, θέλουμε εξαίρεση σχετικά. Και πόσο πόσο σε ποιο βαθμό θα υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις για την ανακύκλωση. Τέλος, για αυτές τις εκτεταμένες σπουδαίες μονάσεις σταθερές και μακρόπνες. Έχει νόημα να, να, να δίνουν τέτοιους χαρακτηρισμούς όταν κάτι το επαναχαρακτηρίζουμε κάθε τετραετία. Αφού είναι κάτι που λέμε να μπορεί να μείνει εκεί 20-30 χρόνια. Όλα αυτά μας είναι απλώς τροχοπέδες, αγρίαστες. Άρα είμαι ανοιχτό σε αυτή τη φάση. Έχουμε κάνα δύο μήνες και τις διακοπές να τα σκεφτούμε και να δούμε τι πραγματικά κίνδυνο θα θεωρηθεί ότι υπάρχει. Και παράταση να δώσουμε, κανένα, καμία αντίρρηση. Να μην μας ε, στριμώξουν γιατί απαγορεύσαμε κάποια πράγματα δίκως. Mm-hmm. Uh, Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την κυρία Εύανς να την ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ καλή έκθεση όπου συμφωνώ σε πολλά σημεία. Ανέφερε ότι ένα ειδικό πρόβλημα υπάρχει στην ε, επεξεργασία των αποβλήτων των παλαιών ε, συσκευών όπου εμπεριέχονται αλογονούχα, PVC, και άλλες επικίνδυνες ουσίες και με την θερμική αντιμετώπιση τέτοιων αποβλήτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τρίτου Κόσμου κατά την αποτέφρωση δημιουργούνται φουράνια και διοξίνες. Και είπε ότι αυτά μόνο με υψηλή θερμοκρασία σε ειδικούς αποτεφρωτές μπορεί αυτό το φαινόμενο δημιουργίας φουρίνων και διοξινών να αποφευθεί. Τώρα, σε σχέση με μελέτες παγκόσμια, είδαμε ότι τα παιδιά στα παιδιά σημειώνεται υψηλότερη περιεκτικότητα διοξίνης στο αίμα τους από ό,τι στις μητέρες τους. Ιδιαίτερα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, που τα απόβλητα σε χωματερές ε, τα παίρνουν και προσπαθούν να τα πουλήσουν. Και ακόμα και στην θάλασσα και ε, ανακαλύπτονται υπολείμματα διοξίνης. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Εύανς για την διάσκεψη για αυτό το θέμα και την ακρόαση με οι δήμονες πολλά στοιχεία μπορέσαμε να αποκομίσουμε από αυτή την ακρόαση. Και τώρα με την οδηγία ΡΟΣ, εκείνο περί του οποίου πρόκειται είναι το περιβάλλον και τους ανθρώπους από διαρκείς βλαπτικές επιπτώσεις από τέτοιες ουσίες να τους προστατέψουμε. Εδώ πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούμε για την αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών στην παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Και κάποιες ουσίες δεν επιτρέπεται καθόλου στην παραγωγή να χρησιμοποιούνται πια πιστεύω εγώ, όπως ε, τα διφενήλια και όπως άλλα χλωριούχα, χλωριούχες ουσίες ε, ε, όπως το κάδμιο το, και ο μόλιβδος και ο υδράργυρος. Νομοθετική δηλαδή απαγόρευση σε σχέση με την οδηγία ΡΟΣ και για την χρήση επικίνδυνων ουσιών. Και συμφωνώ και με την κυρία Evans ότι ο κατάλογος απαγόρευσης για επικίνδυνες ουσίες στο, στις παλαιές συσκευές ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρονικών συσκευών δεν μπορεί να είναι ένας κλειστός κατάλογος, πρέπει να είναι ένας ανοιχτός κατάλογος που θα συμπληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο της επιστήμης και των ερευνών το Κοινοβούλιο πρέπει σε διαδικασία συναπόφασης για την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών να συναποφασίζει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την πρόταση. Εξαιρέσεις, ρυθμίσεις εξαιρέσεις για τις επικίνδυνες ουσίες δεν επιτρέπεται να δικαιολογούνται οικονομικά. Η μετάβαση σε ασφαλείς ουσίες απαιτεί έρευνες αν μια εξαίρεση θα έπρεπε να χορηγηθεί, η χρήση επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει στο τεχνικά εφικτό χαμηλότατο επίπεδο, χαμηλότερο εφικτό επίπεδο να γίνεται. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Evans ότι το REACH και το ROSA αμοιβαία αλληλοσυμπληρώνονται όσον αφορά την χρήση χημικών ουσιών. Γενικά χρειάζονται προθεσμίες και διορίες ώστε όσοι εμπλέκονται να έχουν ένα περιθώριο, ένα πλαίσιο ασφάλειας και για την σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Οι εθελοντικές προσπάθειες κάποιων παραγωγών πρέπει με σαφείς ρυθμίσεις ε, να υποστηρίζονται από πλευράς του νομοθέτη ώστε στρεβλές συνθήκες ανταγωνισμού να αποφεύγονται η προστασία περιβάλλοντος δεν μπορεί να επαφείται μόνο και αποκλειστικά στην αγορά, στους παράγοντες της αγοράς. Είναι σκόπιμο να γίνει μια μελέτη ε, για τη μελέτη αντίκτυπου ε, των επιπτώσεων της οδηγίας ΡΟΣ, ώστε τα αποτελέσματα έγκαιρα να εξεταστούν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να αξιολογηθούν και να λυθούν υπόψη από αυτήν. Και τέλος θα ήθελα να προτείνω και να πω ότι σκόπιμο θα ήταν η σωστή απόφαση του Κοινοβουλίου για την οδηγία Ρώσο να συνδεθεί με την εκστρατεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την απαγόρευση των PVC. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ρίχαρτ Βέμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω, ως θέμα αρχής, θα, θα έπρεπε σε σχέση με τη διαδικασία recast για την ε, αναδιατύπωση αυτής της ε, οδηγίας ε, κανονικά θα έπρεπε μια νέα πρόταση να υποβληθεί και όχι να έχει γίνει recast αναδιατύπωση. Συμφωνώ με τους συναδέλφους σε σχέση με το Ρώσα και το Rich μια και αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται και για την επέκταση του καταλόγου που θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για την πρόσθεση νέων ουσιών. Τώρα, όσον αφορά τι προτάσει τη για το σωστό συσχετισμό με το REACH δεν σύμφωνο απόλυτα, Γιατί με το REACH έχουμε μια διεργασία, μια διαδικασία που δημιουργήσαμε που ανταποκρίνεται πολύ καλά στις ανάγκες και απαιτήσεις του πληθυσμού για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν μπορούμε να δούμε πώς εδώ σε ένα ξεχωριστό τομέα για τα ηλεκτρονικά και τις ηλεκτρικές συσκευές ε, να χρησιμοποιούμε ένα ξεχωριστό τομέα και βλέποντας τις δυνατότητες του REACH ε, που υπάρχουν για αυτή την ομάδα προϊόντων και την ε, πραγματογνωμοσύνη των επιστημόνων όσον αφορά τις διεργασίες REACH, ε, θα μπορούσαμε ιδιαίτερα οι ουσίες που προαναφέρθηκαν και οι διατάξεις να είναι επικοδομητικές ώστε να μπορέσουμε να μεταθέσουμε αυτές τις διαδικασίες για να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα, στα σωστά αποτελέσματα και όσον αφορά τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτή η, σε τακτά διαστήματα επανεξέταση και όσον αφορά την ε, τις εξαιρέσεις, τις άδειες εξαιρέσεων ή την εκνοή τους. Νομίζω δεν ανταποκρινόμαστε απόλυτα στην ε, οικονομική πραγματικότητα και στις ανάγκες αυτής της πραγματικότητας υπάρχει εδώ και το θέμα της ε, μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών ε, και για την ανάλυση αυτή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η ίδια η πραγματικότητα θα έλεγα δεν βαίνει πάντα εκ παραλίλου με το ευχολόγιο που θέλουν να υλοποιήσουν κάποιοι συνάδελφοι. Και θα ήθελα να πω ότι σε αυτόν τον τομέα η προστασία των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά και το εφικτό και το δυνατό του να επιτευθούν οι στόχοι υπέρ των καταναλωτών είναι σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν σε σχέση με τις σκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μην έχουμε αποδυναμώσει, να μην αποδυναμώσουμε με κανένα τρόπο αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε πολλαπλά. Θα ήθελε να ανταποκριθεί. Ποιος θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Που είναι... Πολύ Έχει πάρα πολλά σχόλια και πολύτιμες πληροφορίες. Θα διατρέξω τα βασικά σημεία που ακούστηκαν σήμερα το βράδυ. Ορισμένα από αυτά τα έχω αναφέρει ήδη σε προηγούμενες συζητήσεις. Ε, αν τα έχω επαναλάβει, ε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά τα ίδια ερωτήματα προέκυψαν και τώρα. Θα ξεκινήσω με το πεδίο εφαρμογή. Όπως εξηγήθηκε ήδη, όταν η Κομισιόν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, είχαμε λάβει σαφή εντολή να απλουστεύσουμε σαφώς και να καταστήσουμε πιο απλή και πιο σωστά εφαρμοστέα την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, δεν μελετήσαμε την επίπτωση που θα έχει μια ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Αναφέρθηκε επίσης ότι αναφύεται μια συνένεση για την παρέκταση του πεδίου εφαρμογής. Μάλιστα μίλησαν ορισμένοι για ένα ανοιχτό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ε, αυτή η συνένεση δεν εμπεριέχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας το λέω από τώρα για τους εξή λόγους. Δεν θέλουμε να κάνουμε νομοθετική πρόταση. Ε, χωρίς να έχουμε μελετήσει την επίπτωση. Δεν έχουμε ιδέα ποια επιπλέον προϊόντα θα πρέπει να προσθεθούν, δεν έχουμε ιδέα τι υποκατάστατα θα πρέπει να ε, υπάρξουν, για ποια προϊόντα θα πρέπει να υπάρξουν ε, υποκατάστατα, πόσο ασφαλή είναι, πόσο αξιόπιστα είναι. Επομένως, προς το παρόν, η Κομισιόν ε, είναι διστακτική στο να συμφωνήσει με ένα ανοιχτό πεδίο χωρίς ε, μελέτη αντικτύπου. Όπως σας είπαμε και σε προηγούμενες ε, συνεδριάσεις, ε, παρότι έχει ακουστεί αυτό το ανοιχτό πεδίο, εμείς δεν το βλέπουμε εφικτό. Για το θέμα του ΡΟΣ σε αντιδιαστολή με το ΡΙΤΣ. Αντίθετα με το πρώτο σημείο, εδώ συμφωνούμε με αυτά που είπε η συγγήτρια. Πιστεύουμε ότι το ΡΙΤΣ και το ΡΟΣ είναι συμπληρωματικά νομοθετήματα και συνυπάρχουν και συμπληρώνουν το ένα το άλλο, θαυμάσια. Επίσης, ε, εδώ η αναφιόμενη αυτή η συνένεση συμπεριλαμβάνει και την Κομισιόν. Τώρα, οι νέες ουσίες, δύσκολο θέμα αυτό. να μην ξεχνάτε και κάποια υποθέματα. Δηλαδή, το θέμα ποιες χημικές ουσίες, πώς θα τις προσδιορίσουμε και πώς θα τις ε, εντάξουμε σε κάποια νομοθετήματα. Υπάρχουν τρία υποθέματα, λοιπόν, λοιπόν εδώ κάποιε κάποιες φορές τα μπερδεύουμε. Καταρχάς, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του πώς καθορίζουμε ποιες ουσίες πρέπει ή θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην νομοθεσία. Γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε συμπεφωνημένη μεθοδολογία. Ούτε εμείς, ε, η Κομισιόν, ούτε το νομοθετικό σώμα έχει μια σαφή μεθοδολογία για το πώς αποφασίζουμε αν μια ουσία θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να προσθεθεί στον κατάλογο. Και αυτό είναι ένα κενό που η παρούσα πρόταση της ε, Κομισιόν θα ήθελε και προσπαθεί να καλύψει. Προτείνουμε με κάποιο τρόπο, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, προτείνουμε πάντως να δημιουργήσουμε από κοινού μια συμπεφωνημένη και σαφή μεθοδολογία, μεθοδολογία ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το πώς αποφασίζουμε ε, το ποια υποκατάστατα, το ποιες ουσίες θα συμπεριληφθούν ή όχι. Η μεθοδολογία λοιπόν δεν ισοδυναμεί ε, τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι πώς εντάσσουμε την ε, μεθοδολογία στα πλαίσια του νομοθετήματος. Πώς την κάνουμε νομοθεσία. Και τώρα, θα πρέπει ως διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε τη συναπόφαση ή θα ήταν πιο πλεονεκτικό να χρησιμοποιήσουμε ως διαδικασία την ε, επιτροπολογία δηλαδή να δοθεί εντολή στα πλαίσια επιτροπολογία στην Κομισιόν να κάνει προτάσει. Εμεί σα προτείναμε την επιτροπολογία για διάφορου λόγους θετικούς κατά την άποψή μας προφανώ, Καταρχάς, μια τέτοια διαδικασία εντάσσεται σωστά και μπορεί να δώσει γρήγορα αποτελέσματα, πιο γρήγορα από τη συναπόφαση. Επίσης, μπορεί να δώσει αποτελέσματα ε, πιο στοχευμένα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε διαθεσμικές συμφωνίες για να θεωρήσεις Με πολύ συγκεκριμένο και εστιασμένο τρόπο θα αλλάξουμε συγκεκριμένες ουσίες και δεν θα πειράξουμε τίποτε άλλο. Και επιπλέον, όπως είπα και προηγουμένως, θα λειτουργεί με βάση ε, μία σαφή μεθοδολογία, με μία σαφώς προσδιορισμένη μεθοδολογία. Επίσης θα είχε και ένα άλλο πλεονέκτημα. Θα έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους ε, ε, εμπορευόμενους, στους ε, οικονομικούς φορείς, στους διοικητικούς παράγοντες, γιατί είναι η διαδικασία συναπόφασης, όπως αυτή που πρότεινε η συγγήτρια, με αναθεώρηση κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει. Μια μόνιμη εξέταση της οδηγίας. Μόλις αποφασίσουμε τη μία εκδοχή της οδηγίας θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και θα ακολουθήσει μια νέα ε, πολιετής ε, τέτοια διαδικασία στην απόφαση. Δεν είναι ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε και να συσσωρεύσουμε εξουσίες. Ε, δώστε μας μια τέτοια εντολή επιτροπολογίας για πρακτικούς λόγους μόνο. Τρίτο υποσημείο. Ποιε νέε ουσίες θα πρέπει να προσθεθούν. όπω είπα ήδη, σε αυτή τη φάση δεν έχουμε συμφωνήσει για μια μεθοδολογία. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Η Κομισιόν χρησιμοποιεί την παραδοσιακή λογική της να ξεκινάει μια μελέτη, να παραγγείλει μια μελέτη, εξωτερική μελέτη, για να λάβουμε για να συγκεντρώσουμε στοιχεία και να μας δοθούν συμβουλές και υποδείξεις για αυτό το θέμα. Και εδώ η επιχειρηματολογία απομακρύνεται από, το, από τη διαδικασία όπως πραγματικά συμβαίνει. Το γεγονός ότι η Κομισιόν παρήγγειλε μία μελέτη και την πλήρωσε, φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν έχει α, αποποιηθεί και των δικαιωμάτων της ε, υποβολής ε, προτάσεων. Όχι. Παραγγείλαμε την μελέτη, θα πάρουμε τα αποτελέσματα για την ε, μελέτη που πληρώσαμε. Είναι συμβουλές αυτές που θα μας δοθούν, που θα τις λάβουμε υπόψη, αλλά δεν μας υπαγορεύουν το νομοθέτημα που θα προκύψει από εκεί. Η έκθεση που μας παρουσιάστηκε αναφέρει σε πολλά σημεία ότι οι συντάκτες αυτής της μελέτης συνέστησαν το α ή το β. Και αν δείτε το κείμενο θα διαπιστώσετε ότι όντως λέγεται αυτό. Αλλά όμως, αυτό είναι το καθήκον της Κομισιόν. Αν ε, αξιολογήσουμε ισορροπημένα, σωστά αυτή τη μελέτη, διαμορφώνουμε μια διαφορετική εικόνα. Σας παραθέτω, η μελέτη λέει ότι για τις περισσότερες ουσίες για τις οποίες μιλούσαμε σήμερα και προηγουμένως, ε, τα δεδομένα είναι παρκή. Ή οι συστάσεις που κάνει η μελέτη λένε οι συντάκτε ότι δεν είναι επαρκώ βάσιμα ή σε ορισμένε περιπτώσει δεν συνιστάται καμία δράση. Να μην σα κουράσω, αλλά έχω ένα κατάλογο για τους βρωμιούχου ε, φλόγας φλόγα, ε, για το PVC, για τα χλωρινούχα ω πλαστικοποιητέ για μια σειρά από χημικές ενός που δεν μπορώ καν να προφέρω και για μια σειρά από ανόργανες ουσίες, ε, αρσενικό κτλ. Για όλες αυτές τις ουσίες αναφέρονται στην έκθεση προσοχή, λένε οι συντάκτες της έκθεσης. Προσέξτε. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν είναι προσεκτική. Ε, ίσως έτσι εξηγείται το θέμα που, και απαντάτε το ερώτημα που θέσατε, γιατί δεν ε, ακολουθεί τη συμβολή των συντακτών ε, της ε, μελέτης. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία τώρα τον, των λόγων ή μάλλον των παρασκευαστών που έχουν περάσει σε νέες ουσίες, στη χρήση νέων ουσιών. Από μόνοι τους. Κανένα πρόβλημα εάν οι νέε ουσίε παρουσιάζουν ε, καλύτερη περιβαλλοντική προστασία και καλύτερη προστασία τη υγεία. Κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό και μπορούμε να σα ακούσουμε. Ένα ερωτηματικό. Αν αυτοί οι κατασκευαστέ έχουν αξιολογήσει όλες τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία που συνδέονται με τα υποκατάστατα που χρησιμοποιούν τώρα. Γιατί εμείς αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πριν λάβουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Για να προτείνουμε κάτι, μια νομοθεσία για την Ευρώπη. Αυτοί οι κατασκευαστές λοιπόν έχουν, κάνει τέτοια, έχουν λάβει υπόψη τους αυτά τα στοιχεία ε, για τα υποκατάστατα που χρησιμοποιούν. Προσοχή. Όπως και αλλού. Και εδώ προσοχή να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου το φάρμακο είναι χειρότερο από την αρρώστια. Το θέμα της ε, χρήσης ή όχι των ε, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων όταν ε, αποφασίζουμε για τις προσωρινές εξαιρέσεις. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει και προηγουμένως. Εμείς ως Κομισιόν είμαστε πεπισμένοι ότι, είναι κάτι, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Είναι εκ των όνων στη σημερινή πολιτική, στην περιβαλλοντική πολιτική, Αν θέλουμε την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, που τη θέλουμε όλοι μας, ε, βασίζεται αυτή σε τρεις πυλώνες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τους τρεις πυλώνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο και μόνο για λόγους κόστους θα δώσουμε οποιασδήποτε εξαιρέσεις. Όχι. Ούτως ή άλλως δεν θα το κάνουμε μόνοι μας, θα εμπλακείτε κι εσείς. Ακόμη και εσείς στην Επιτροπολογία θα εμπλακείτε με τα δικαιώματα ελέγχου που έχετε αλλά θα πρέπει τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη. Ούτω ή άλλω, εσεί ε, πολλέ φορέ στην Επιτροπή σα ζητάτε να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα να, του να λαμβάνουμε υπόψη το αν οι ουσίε είναι επικίνδυνε ή αν προκαλούν κίνδυνο. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Πιστεύουμε ότι η ΡΟΣ βασίζεται στο πόσο επικίνδυνες είναι οι ουσίες. Αλλά πιστεύουμε ότι η ευθυγράμμιση της κοινωνικής νομοθεσίας, εδώ παραπέμπω στο ΡΙΤΣ βέβαια, η ευθυγράμμιση είναι απαραίτητη και το ΡΙΤΣ βασίζεται στον κίνδυνο που δημιουργείται. Και επομένως μια μελλοντική μεθοδολογία της οδηγίας ΡΟΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το στοιχείο του κινδύνου, του risk. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες και τις πιο κύριες ερωτήσεις. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας, εάν έχετε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, επεξηγήσεις. Ένας έχει ζητήσει τον λόγο, πρώτου εισηγείται δηλαδή τον λόγο, ο κύριος Ταντέους, παρακαλώ. Ε, ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγες παρατηρήσεις έχω. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο που επετέλεσε. Είναι γεγονός ότι έχουμε πολλές απαντήσεις, πολλές προτάσεις, αλλά απομένουν και έχουμε κάποια ερωτήματα. Ας σας αναφέρω σχετικά μερικά. Πρώτον, υποστηρίζουμε την άποψη της εισηγήτριας να αλλάξει το εύρος, το πεδίο της οδηγίας να είναι ένα ευρύτερο, πιο ανοιχτό πλαίσιο. Δεν είμαι όμως σίγουρος αν δίνει επαρκή σαφήνεια και αν θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε χρονοβόρες διαδικασίες ε, και συζητήσεις όσον αφορά ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί. Δεύτερον, δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι αν καταλήγοντας ε, στο ε, κύκλο ζωής των ιατρικών συσκευών θα έπρεπε αυτές να συμπεριληφθούν. Είναι πολύ μακρύς ο κύκλος ζωής ε, για να ε, εντάσσεται εδώ σε σχέση με την παραγωγή μικρού όγκου ε, υλικών. Γι' αυτό κάποια, κάποιες συσκευές συσκεύη δεν θα συμπεριλαμβανόντουσαν. Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει περισσότερα στοιχεία. Δεύτερον, όσον αφορά την εξαίρεση κάποιων συσκευών, απέρευσε από αυτή τη συζήτηση ότι υπάρχει ερωτηματικό αν η περίοδος η τετραετής είναι επαρκής ε, για τις εταιρείες. Έχουμε διαφορετικού τύπου συσκευές ε, σε σχέση με αυτή την οδηγία. Έχουμε ηλιακά πάνελ, όλα πάνελ και κινητά τηλέφωνα πρέπει να συμπεριληφθούν διάφοροι παράγοντες. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων απαιτεί κτλ. Γι' αυτό η τετραετία σε αυτή η περίοδος φαίνεται ότι είναι πολύ σύντομη. Ίσως υπάρχει εδώ κάποιο ερωτηματικό και πρέπει να παραταθεί αυτός ο κύκλος ζωής αυτή η περίοδο. Η κυρία Συγκίτρια λέει ότι ίσως ε, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα. Θα θέλαμε όμως να δοθούν συγκεκριμένες επεξηγήσεις σε ποιε περιπτώσεις και πώς αυτές οι εξαιρεσει θα θεσπίζονται και θα δίνουν Τέταρτον, κάποιες ουσίες ε, υπάρχουν που θέλει να απαγορευτούν η συγγήτρια. Τώρα θα είναι πιο δύσκολο να υποστηριχθεί αυτό παρότι έχουν παρουσιαστεί κάποια επιχειρήματα και τεκμήρια. Είναι αρκετά επιλεκτική όμως αυτή η διαδικασία και δεν είναι απόλυτα δικαιολογημένη για τόσο ριζοσπαστικούς περιορισμούς γνωρίζουμε και από άλλες αναλύσεις ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με κάποια στοιχεία που παρουσιάζονται και από πλευρά τη έκθεση. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει η μία ενιαία σαφής μεθοδολογία. Γι' αυτό δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη η έκθεση αυτή και δεν θα είναι δυνατόν απόλυτα να την υποστηρίξουμε μέριστα. Κατανοούμε γιατί η συγκίτρια δεν θέλει να ληφθούν οι αποφάσεις σε διαδικασία επιτροπολογίας. Μια και όμως αυτά τα θέματα είναι τόσο περίπλοκα και τόσο σύνθετα θα έπρεπε να υπήρχε μια διαδικασία επιτροπολογίας με εποπτεία, με έλεγχο εποπτευόμενη. Θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτηση εναλλακτικών τέτοιων ουσιών. Εκτιμούμε και θεωρούμε ότι κάποιες επιχειρήσεις υιοθετούν τη μέθοδο των πρακτικών, Όμω οι δικέ του λύσει όπω υιοθετούνται μπορεί να μην είναι οι πιο ενδεδειγμένες και οι καλύτερε για τι υπόλοιπε επιχείρησει. Έχουμε και μία ακόμα επιφύλαξη, Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Πρέπει να επαρκεστώ σε αυτόν τον χρόνο που μου δώσατε και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Το τελευταίο είναι το PVC. Δεν είναι απόλυτα σαφέ αυτό για μας. Δεν είναι απόλυτα σαφέ αν η απαγόρευση των PVC είναι η βέλτιστη, η καλύτερη μέθοδος. Η κυρία εισηγήτρια έχει μια στεναρότατη άποψη για αυτό το ζήτημα, όμως δεν έχει αναφέρει τις, ε, α το πω έτσι, ουσιοδέστερες ε, ε, αλλαγές όσον αφορά την διαδικασία ΡΟΣ. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε πολύ καλά να επιληθεί εκτός αυτής της οδηγίας. Τα προβλήματα σε σχέση με αυτό το θέμα μπορούν έτσι να επιληθούν και όχι απαγορεύοντας κάποιες ουσίες ή προϊόντα. Επίσης αν θέλουμε να περιορίσουμε την χρήση των PVC που χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα και σε πολλούς τομείς ε, βιομηχανιών όπου εξαρτώνται θέσεις απασχόλησης από αυτές τις μεθόδους παραγωγής, θα πρέπει να σκεφτούμε τις οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσεις αυτής της απόφασης. Αν, να, αν αποφασιστεί να ενταχθεί το PVC στο πλαίσιο ε, του πεδίου οδηγίας, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να λάβουν υπόψη αυτά που είπα για σαφή μεθοδολογία επιστημονική που πρέπει να υιοθετείτε όταν ε, επιβάλλουμε νέους περιορισμούς. Ευχαριστώ. Yeah, Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιμάνσκι. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και όλους τους αδέλφους αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι δελεχός και με θετικό πνεύμα μας είπαν τις παρατηρήσεις τους. Ξέρω τώρα ότι πιέζει ο χρόνος και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση. Αλλά κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να ξαναλύσουμε αυτή την οδηγία, οπότε και θα μπορέσουμε, ελπίζω, να ξανά έχουμε την ευκαιρία. Τελικά Όλα αυτά να τα συζητήσουμε πιο λεπτομερώς τώρα. Κάτι για τη διαδικασία και ξεκινάμε πρώτα-πρώτα με την ε, προθεσμία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτως ώστε να παραταθεί η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Όμως, όμως, να διατηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν περιθώρια. Ξέρω ότι για την οδηγία δεν έχετε όλοι τα κείμενα. Παράλληλα προχωρήσαμε, γι' αυτό και υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Ε, ξέρω ότι ο έχει πρόβλημα με την οδηγία ΡΟΣ. Ελπίζω τελικά να μην έχετε πρόβλημα, να πούμε να προχωρήσουμε παράλληλα τα δύο νομοθετήματα. Γιατί δεν μπορεί μία υποχρέωση να μην την άλλη. Τώρα. Όντω, κάποιοι προτιμούν την επιτροπολογία, κάποιοι την συναπόφαση και σε σχέση με το πεδίο τώρα όσον αφορά αυτούς τους θερμοσορευτές Υπήρξε μεγάλη πίεση από κάποια εταιρεία. Και τελικά αποφάσισα να υπάρξει μια παρέκκληση στη ρύθμιση, αλλά όχι απόλυτη εξαίρεση. Το κύριο Σόνικ, ότι 3,5 χρόνια είναι λίγα για σταδιακές καταργήσεις. και τους υπερβραδιντές και το PVC. Εδώ για μια δεκαετία δεν συζητάμε. Και από το 2003 η βιομηχανία επεξεργάζεται λύσεις. Και όσοι από εσά πριν από λίγες μέρες παρέσετε σε εκείνο το σεμινάριο ακούστηκαν απίστευτα πολλές πληροφορίες. Από πλευρά Apple, πλευράς Nokia και άλλων εταιριών μας είπαν όχι μόνο πώς γίνεται αυτό, αλλά και πώς βοηθήσαν και τις μικρότερες εταιρείες σε όλη την αλυσίδα της ε, παραγωγής, της προσφοράς. Σε σχέση με τις ΜΜΕ εξετάστηκε τι χρησιμοτοδοτήσεις είναι ε, εφικτές. Όλα αυτά τα είπαμε στο σεμινάριο. Άρα, είπαμε ότι αν οι εταιρείε μπορούν να βρουν υποκατάστατε συσκευέ, προϊόντα, τότε μπορούν να τύχουν εξαίρεση. Και φοβάστε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να έχουν πρόβλημα αυτέ οι τόσο πρωτοπόρε, τόσο μεγάλε εταιρείε να μην μπορούν να βρουν κάποιε αξιόπιστε λύσει. Το είπε και η Κομισιόν. Για τι υποκατάστατε ε, συσκευές και προϊόντα. τα bioaccumulative, τα ότι μπορεί και να είναι πιο αποδοτικά από τα αρχικά προϊόντα. Πάντως βεβαίως και κρεμούν ακόμα πολλά που θα πρέπει να τα συζητήσουμε να τα διερευνήσουμε σε συνεργασία με τους και ηγητές. Θα συνεχιστεί ο προβληματισμός μας. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ähm, äh, σε ευχαριστούμε και το αίτημα αυτό για το ΡΟΣ να μπορέσει να ενταχθεί και ταυτόχρονα στην Ολομέλεια να μπορέσει να εξεταστεί έτσι στον κύριο Φλόρεντ πρέπει να το πούμε και να συζητήσουμε μαζί του να προαγάγει την έκθεση αυτή και να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Τώρα θα προτείναμε, θα λέγαμε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών η 24η Φεβρουαρίου. Θα επεκταθεί, όχι 14 Ιανουαρίου, 24 Φεβρουαρίου, εντάξει. Συμφωνείτε, 24 Φεβρουαρίου. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την έκθεση κοντά σε αυτή την προθεσμία με τις τροπολογίες και τα λοιπά. Ωραία. Και ολοκληρώσαμε τη σημερινή συνεδρία. Σε ευχαριστώ που συμμετείχατε. Αύριο θα τα πούμε στις 10 η ώρα. 10 η ώρα θα συνεχίσουμε. Για τους συντονιστές στις